Συνάδελφοι, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, ξέρετε προφανώς ότι το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση αυτής. Αναγνώριση του Προέδρου. Το πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το απόγευμα είναι η συζήτηση για τις προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και δεν θα υπήρχε καλύτερο τρόπο να συζητήσουμε τι προτεραιότητε τη Επιτροπή μα με τόσου λίγου ε, ευρωβουλευτές παρόντες ε, στη συνάντηση. Με αυτούς τους λίγους λοιπόν που είμαστε εδώ θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αλλαγή στην εμίσια διάταξη. Η Τάνια Φαγιόν, η συνάδελφος, ζήτησε εν ώψη της ψηφοφορία που θα γίνει τη Δευτέρα για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο να ε, προσθεθεί στις ψηφοφορίες. Υπάρχουν αντιρρήσεις, η κυρία Ίντβελτ. Όχι, δεν έχω αντίρρηση στην αλλαγή. Όμως με μπερδεύει λίγο αυτό το πρώτο σημείο της μερικής διάταξης για το οποίο έχετε αφιερώσει, προβλέψει δύο ώρες. Δύο ώρες για τις προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ παρακολούθησε απόφαση των συντονιστών της 11ης Ιουλίου 2019. Εγώ ήμουν σε εκείνη τη συνεδρίαση, αλλά ε, έχω μια πολύ διαφορετική ανάγνωση της απόφασης. Δεν ξέρω τι ακριβώς συζήτηση πρόκειται να κάνουμε, ούτε ποιο θα είναι το συμπέρασμα αυτής της συζήτησης. Έχουμε όλοι τις προτεραιότητες των πολιτικών μας ε, ομάδων, θα γίνουν οι ακροάσεις με τους επιτρόπους, η επιτροπή μετά θα ε, παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών τη και μετά μπορεί να συζητήσουμε και για τις προτεραιότητες. καταλαβαίνω τι, τι, τι είδους ε, συζήτηση θα γίνει σήμερα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό το σημείο στη μέρη διάταξη. Πρόεδρο. εντάξει, καταλαβαίνω τη θέση σα, αλλά οι συντονιστέ ήταν όλοι παρόντες και είχαμε πει ότι θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να προβλέψουμε ποια θα είναι η κατάσταση ε, εν ώψη των ακροάσεων που θα γίνουν με τους οριστέντες επιτρόπους και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έτσι είπαν και οι συντονιστές ε, να συζητηθούν τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Λίμπε. Κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ. Παρά το γεγονό ότι καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση για τι προτεραιότητε, στην ουσία προετοιμαζόμαστε για τι ε, ακροάσει των ε, επιτρόπων. Και όλε οι πολιτικέ ομάδε αυτό κάνουν στην ουσία. Και κοιτάζοντα στην, ε, στην αίθουσα, Αναρωτιέμαι, θα τις καθορίσουμε σήμερα τις ε, προτεραιότητες Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Εδώ λείπουν ακόμη και ορισμένοι συντονιστές από την ε, συνεδρίαση. Γεια σας κύριε Λένας, είστε και ένας από τους συντονιστές. Σας καλωσορίζω. Ωραία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έλεγα, γιατί το ενδιαφέρον που εκφράζεται για αυτή τη συζήτηση είναι τόσο χαμηλό και τι συμπέρασμα βγάζουμε Λαμβάνοντα υπόψη ακριβώς τον πολύ μικρό αριθμό συναδέλφων που βρίσκονται σήμερα εδώ στην αίθουσα. κυρία Βέντκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά, προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει αυτή η συζήτηση. Όμως το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι τι θα γίνει με τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Γιατί θα υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στα θέματα που θα θέλουν κάποιοι να ιεραρχήσουν ε, ως θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν, να απασχολήσουν τη ΛΥΜΠΕ. Αλλά δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Ε, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση εμεί εδώ. Θα πρέπει το θέμα να αναπευθεί και πάλι στου συντονιστέ. Οπότε μπορείτε να μα πείτε λίγο τι ακριβώ θα γίνει σήμερα, αυτά στα οποία θα καταλήξουμε, τι θα τα κάνουμε μετά και πώ θα πάμε στου συντονιστέ. Πρόεδρο, συμφωνώ ακριβώ με αυτό που λέτε. Το είπα και λίγο ηρωνικά ξέρετε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είναι τρίτη, εν πάση περιπτώσει, σε τελική ανάλυση. Δεν είναι Παρασκευή βράδυ, τρίτη είναι ακόμη. Οπότε έχουμε τακτική συνάντηση, συνεδρίαση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Βεβαίως τα μέλη οφείλουν να είναι εδώ και ξέρετε, γι' αυτό ξεκίνησα και με, αυτό το ειρωνικό σχόλιο, γιατί βλέπω ότι είναι πράγματι πολύ λίγοι αυτοί που προσήλθαν στη συνεδρίαση, οπότε μπορούμε ίσως να ε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση εντάχει, αν θέλετε, και να επικεντρωθούμε ταυτόχρονα και στην, ε, ε, στην προετοιμασία των ακροάσεων που θα γίνουν στο τέλος του μήνα, από το τέλος του μήνα και στη συνέχεια ε, γιατί αυτό είναι το βασικότερο θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αν εσείς τώρα έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένα, κανένας λόγος να έχουμε αυτό το θέμα στη μύρια διάταξη, μπορούμε να το, να το αφαιρέσουμε και να γίνει η σχετική συζήτηση, η αντίστοιχη συζήτηση, αύριο στους συνείδρες των συντονιστών. Η κυρία Έντβελτ. Ναι, νομίζω ότι θα είχε νόημα αυτό, διότι όσον αφορά τις ε, ακροάσεις, έχουμε ήδη καθορίσει τι προτεραιότητε τη Επιτροπής μα στι γραπτέ ερωτήσει που έχουμε αποστείλει στους Επιτρόπους. Στη συνέχεια οι προ... προφορικές ερωτήσεις εξαρτώνται, επαφίονται στις ε, ε, πολιτικέ ομάδε και στου μεμονωμένου ευρωβουλευτέ. Δεν θα αποφασίσουμε εμεί εδώ. Δεν πρόκειται να πάρουμε κάποια απόφαση σχετικά με κάποιο πρόγραμμα εργασιών. Οπότε πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι θα συζητήσουμε και τι θα αποφασίσουμε. Όπω είπε και η συνάδελφο, πολύ σωστά, ίσως θα μπορούσαμε το χρόνο που έχουμε να τον αξιοποιήσουμε καλύτερα. Πρόεδρος, ωραία. Να σας πω κάτι όμως, στις ανακοινώσεις του Προέδρου ε, δεν σηκώσατε τα χέρι, το χέρι σας, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο. Φαίνεται όμως ότι ήδη υπάρχει μια διαφωνία για το αν θα έχει νόημα να γίνει αυτή η συζήτηση σε τακτική συνεδρία της, ομάδας, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και παράλογο να θέσει ένα τέτοιο θέμα τρίτη απόγευμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Ε, δεν θα ήταν και ε, τόσο περίεργο να αποφασίσει η Επιτροπή Λίμπη ότι θέλει να τα συζητήσει αυτά τα θέματα, αυτό το θέμα συγκεκριμένα. Αλλά δώσω το λόγο στον κύριο Τζέλο πρωτού περάσω στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Εντάξει, ας ε, μην υπερβάλλουμε. Καταλαβαίνω ότι εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το μικρό αριθμό ευρωβουλευτών που βρίσκονται εδώ. Όμως το ΕΛΚ ήταν μία από τις ομάδες που υποστήριξε να γίνει αυτή η συζήτηση Ακριβώ γιατί είμαστε και μια επιτροπή όπου υπάρχουν πολλά νέα μέλη και θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να γίνει μια τέτοια συζήτηση εκ των προτέρων προτού περάσουμε στους επιμέρους, ε, στα, στα επιμέρους χαρτοφυλάκια για να γίνει και μια ανταλλαγή απόψεων για το ποιε θα είναι οι προτεραιότητε μα για τα επόμενα χρόνια. Φυσικά ε, οι ακροάσει είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά δεν είναι η μοναδική. Επίση, δεν θα μπορούν όλοι να παρίστανται στι ακροάσει. Το να γίνει λοιπόν αυτή η συζήτηση θεωρούμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να ακουστούν οι απόψει όλων εκείνων που θέλουν να, να συμβάλλουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη συζήτηση αυτή. Α ε, επικεντρωθούμε λοιπόν καλύτερα στην ποιότητα των συνεισφορών και όχι στην ποσότητα, δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην γίνει συζήτηση. Πρόεδρος, βλέπω ότι υπάρχει έδαφος σύγκλησης μεταξύ των θέσεων που μόλις εκφράστηκαν και μεταξύ της θέσης που εξέφρασε η κυρία Ζίπελ που εκπροσωπεί του σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Υπάρχουν ευρωβουλευτέ αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, οπότε μπορούμε τουλάχιστον να επιχειρήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση. Αλλά θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον να κάνω τι ανακοινώσει γιατι γιατί πρωτού καλά-καλά ξεκινήσουμε, δεν είχα και την ευκαιρία να ξεκινήσω με, το, με το, τα βασικά, τα, τα συνήθη. Διερμηνία, ξέρετε, τα γνωστά. Όλε οι γλώσσε, εκτό από Ιρλανδικά, ψηφοφορίες θα γίνουν με ηλεκτρονική κάρτα γιατί έχουμε μια σειρά από ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν στις 6 το απόγευμα το βράδυ σήμερα σε λίγες ώρες δηλαδή οπότε σας θυμίζω να έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές σας κάρτες έως εκείνη την ώρα γιατί έχουμε μια σειρά από ψηφοφορίες που πρέπει να κάνουμε και μετά υπάρχει και το επίσης σύνηθες θέμα ε, έγκριση των ε, συστάσεων των αποφάσεων των συντονιστών για τον διορισμό των εισηγητών στα διάφορα θέματα. Ο κ. Λένερς ορίστηκε εισηγητή για τις προϋποθέσεις πρόσβασης ε, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών, το ΕΚΛΙΣ, TCN, και για την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση της πρόσβασης σε ε, άλλων ε, ευρωπαϊκών συστημάτων στο ETIAS. Λένερς όπως είπα. Γιαντβίγκα ε, Βυσνιεύσκα έχει οριστεί η συγγήτρια για το πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας και Λιχτενστάιν όσον αφορά τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τη θέσπιση του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήματος ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία όσον αφορά την πρόσβαση στο Eurodac. Και το αντίστοιχο πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας. Πάλι για τα ίδια θέματα, Eurodac βασικά. Επίσης, ορίστηκε η συγγήτρια η Μαρίνα Καλιουράντ για τη συμφωνία μεταξύ Μεξικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταφορά και την επεξεργασία δεδομένων μητρώου ονομάτων επιβατών. PNR, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεξικό. Κατερίνα Κινίτσι σχετικά με τις διαπραγματε... με... για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την ε, πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Και τα δύο αυτά θέματα στην κυρία Κινίτση. Επίσης, Καρυξοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Στο πλαίσιο του Ταμείου Μετανάστευση και Ασύλου και του Προγράμματος Εργασιών για το 2019, εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε στις 18 Σεπτεμβρίου το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Κομισιόν για την τροποποίηση της ε, εκτελεστικής απόφασης σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μετανάστευση και Ασύλου. Με την παραλαβή αυτού, αυτής της ε, πράξης, της εκτελεστικής, Μάλλον η πράξη αυτή ε, κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω του newsletter στις 19 Σεπτεμβρίου και ορίστηκε και προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Όπως και να έχει, αν υπάρχει κάποιος ευρωβουλευτής που έχει ένσταση, ας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τη γραμματεία ε, της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ έω τι 2 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ωραία, τελειώσαμε και με τις ανακοινώσει. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Σκοπός ήταν να ξεκινήσει... Λοιπόν, ξεκινήσει, ξεκίνησε η κοινοβουλευτική θετία τον Ιούλιο. Έγιναν κάποιες επαφές με όλους τους επιτρόπους, με όλους τους επιτρόπους, τους απερχόμενους επιτρόπους. Τους επιτρόπους της Επιτροπής που ήταν αρμόδιοι για θέματα για τα οποία είμαστε αρμόδιοι και εμείς ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Επίση, έγιναν ακροάσει με όλου του ε, διευθυντέ και επικεφαλεί των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνη, των πολιτικών ελευθεριών και των εσωτερικών υποθέσεων. Είχαμε και συνάντηση συνεδρίαση των συντονιστών στι 11 Ιουλίου, στην οποία αποφασίστηκε να γίνει μια συζήτηση ώστε να δοθεί δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να εκφραστούν, να τοποθετηθούν σχετικά με τις προτεραιότητες για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Μας απομένουν λίγες μέρες έως τις ακροάσει των οριστέντων επιτρόπων. Των επιτρόπων υπό την ε, Επιτροπή της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Και το αντίστοιχο κοινοβουλευτικό έργο που αναμένεται να γίνει στη διάρκεια της θητείας της νέας Επιτροπής και που θα μας απασχολήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα απορροφήσει το περισσότερο χρόνο μας κάποια θέματα, κάποιοι φάκελοι που εκκρεμούν, μάλιστα θα μας ξαναπασχολήσουν και σήμερα στις ψηφοφορίες που θα γίνουν το βράδυ. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ελεύθερα, να τοποθετηθούμε, προκειμένου να συμπληρώσουμε και τη συζήτηση που έγινε στους συντονιστές. Και φυσικά η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο στην ε, αυριανή συνεδρίαση των συντονιστών που θα γίνει το μεσημέρι, το μεσημέρι. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τους συντονιστές και από εκεί και πέρα όποιο μέλος της Επιτροπής θέλει να τοποθετηθεί βεβαίως θα έχει την δυνατότητα να το κάνει και θα καταγράψουμε όλες τις απόψεις που θα ακουστούν. Κύριε Λένερς, έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πιο σημαντικό, πιστεύω, είναι αυτό που μας απασχόλησε και τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, η μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Και αν δείτε τις επιστολές ε, προς τους ε, οριστέντες επιτρόπους και προς την οριστή σε επίτροπο της Επιτροπής, και ε, προς όλους, θα δείτε ότι ε, σαφώς μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και είναι απαραίτητο ένα νέο σύμφωνο. Δεν θα πρέπει να πάει χαμένη όλη η δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε θέματα όπως ε, η Eurodac, παραδείγματος χάρη, που απλώς πρόκειται για μια βελτίωση της καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων των ετούντων άσυλο, παραδείγματος χάρη. Ανεξάρτητα από το τι θα συμφωνηθεί για το Δουβλίνο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να συνεχιστεί. Η αχίλιος πτέρνα λοιπόν της μετανάστευσης αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι το ότι δεν έχουμε αποτελεσματική πολιτική για τις επιστροφές. και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία ε, οι μισοί από αυτούς που θεωρούνται ότι δεν ε, έχουν δικαίωμα ε, προστασίας παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την υποστήριξη από το δημόσιο είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να γίνεται η προστασία των πραγματικών προσφύγων ακόμη και αυτοί που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία, παρατείνουν την παραμονή του και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δικαιολογήσουμε και στην κοινή γνώμη. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε ριζικές ε, αλλαγέ και πρόοδου σε αυτόν τον τομέα, αλλά σαφώς ε, τμήμα τη λύση είναι και η συνεργασία με τρίτες χώρες, ε, χώρε διέλευση, και αυτό έχει κέρια σημασία. Τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. και δεν εννοώ ότι θα πηγαίνει κάθε Υπουργό Εξωτερικών ή κάθε Υπουργό υπεύθυνο για θέματα ασύλου και μετανάστευση από κάθε χώρα στι αντίστοιχε χώρε με τι δικέ του ιδέε, αλλά θέλουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα υποστηρίζεται από όλου του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων και Υπουργού Υπευθύνου για το Άσυλο και τη, Μετανάστευση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, Πρόεδρε, γιατί θέλω να μιλήσω και για την ε, εσωτερική ασφάλεια. Δύο λεπτά μόνο. Ζητώ συγγνώμη γιατί ξεπέρασα το χρόνο μου. Δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής έχει. Πρόεδρος. Είμαστε ακόμη στην προθέρμανση, οπότε σας αφήνω ε, λίγο περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, ε, επεκτείνομαι λίγο και στο θέμα της ασφάλειας. Και στην προηγούμενη θητεία κάναμε πολλή δουλειά για την ασφάλεια και εδώ έχει μεγάλη σημασία η υλοποίηση. Βλέποντας την διαλειτουργικότητα, το αίτιας για το σύστημα αδειοδότησης ταξιδίου, βλέποντας το PNR. Όλα αυτά έχουν το κλειδί τους στην υλοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λένας. Θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να περιοριζόμαστε στα δύο λεπτά ο καθένας. Κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που γεμίζει σιγά σιγά η αίθουσα έρχονται και συντονιστέ για να είναι πιο χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων. Θα προσπαθήσω να μην πάρω πολύ από το χρόνο σας σε αυτή την προκατακτική συζήτηση. Ξεκινώ με μια γενική παρατήρηση. Μιλάμε πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα όμως η ψηφιοποίηση είναι κάτι που καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, στη γεωργία, στις κατασκευές, στην απασχόληση, την ασφάλεια, το ποινικό δίκαιο, την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς επιδρά αυτό στην ατομική συμπεριφορά των πολιτών. Είναι πολύ εύκολο να αγοράσει κανείς ένα εισιτήριο, αλλά είναι ε, και πολύ εύκολο να εξαπλώσει κανείς μια ρητορική μίσους. Θέλουμε λοιπόν παράλληλα με αυτά τα οποία γίνονται να διαφυλάσσουμε και τις δημοκρατικές μας αξίες και να δίνουμε και νέες ευκαιρίες σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον χωρίς να ξεπουλάμε τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη όλων των πολιτών σε αυτές τις πολύπλοκες εξελίξεις που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Για κάποια άλλα θέματα τώρα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, όταν μιλάμε για την ασφάλεια και το ποινικό δίκαιο, η Επιτροπή μας στην επόμενη θητεία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση. Τα τελευταία χρόνια αποφασίσαμε πολλά και στο ποινικό δίκαιο, στην καταπολέμηση της εγκληματικότητα και τη τρομοκρατίας. Αλλά αν δείτε όχι μόνο αυτά που αποφασίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και παλιότερα, Ακόμη πολλά από αυτά που συμφωνήσαμε δεν έχουν υλοποιηθεί στην πράξη. Αν δεν υλοποιούνται λοιπόν τα πράγματα, πώς να εξετάσουμε ένα παραθυράκι αφού δεν έχουμε υλοποιήσει αυτά τα οποία αποφασίσαμε. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή μας να εξετάζει την υλοποίηση και να οθούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να οθούμε τα κράτη-μέλη στην πραγματική υλοποίηση των μέτρων. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να μιλάμε για μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν υλοποιούνται. Τέλος, τελευταίο σημείο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Έγινε πολύ πρόσφατα μία συνάντηση στη Μάλτα και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέρον να τα δούμε. Γιατί μπορεί αυτή η συνάντηση στη Μάλτα να αποτελέσει αφετηρία για να κάνουμε πρόοδο στο να αναλαμβάνουμε ευθύνη για τους ετούντες άσυλο. Ώστε να μην χάνουμε σιγά σιγά αυτά τα οποία είχαμε κερδίσει στο παρελθόν. και να δούμε κατά πόσο μπορούν να ζητούν έσυλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αν δεν μπορούν να πάρουν θεώρηση διαβατηρίου από τη χώρα στην οποία, ε, από την οποία θέλουν να ξεφύγουν από τα βασανιστήρια ε, ε, και την έλλειψη ελευθεριών, η μόνη τους λύση θα είναι να μπουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν για την νόμιμη μετανάστευση και για την απασχόληση και για το άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Σίπελ. Κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπω είπα και πριν, όταν συζητούσαμε την ημερήσια διάταξη, αυτή είναι μια συζήτηση που είναι λίγο αόριστη, πάει προ όλε τι κατευθύνσει. Οι συνάδελφοι Λένερς και Σίπελ που μίλησαν τόνισαν την υλοποίηση. Συμφωνώ μαζί τους. Πρέπει να προσθέσω όμως και την ε, αναγκαστική εκτέλεση. Πρέπει να εκτελέσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών τα οποία ψηφίζουν τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο αφενός και απουσίας ιασδήποτε προσπάθειας όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη, να εκτελέσουμε αυτά τα οποία αποφασίστηκαν, ακόμη και για αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Χρειάζεται μια αξιολόγηση αυτών που έχουμε επιτύχει πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε νέα μέτρα, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχουμε ψηφίσει ένα μακροσκελή κατάλογο μέτρων και δεν έχουμε αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα όλων αυτών, για το κόστος, για το αν χρειάζεται πιθανά αναθεώρηση για κάποια από τα μέτρα αυτά ή και αντικατάσταση. Το άσυλο αναφέρθηκε. Και η νόμιμη μετανάστευση εργαζομένων επίσης είναι ένα θέμα που πρέπει να εξετάσουμε, γιατί αν δεν υπάρχει νόμιμη διέξοδος, δεν θα υπάρξει και λύση στο πρόβλημα του ασύλου. Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμένη στις προστασίες δεδομένων, στον τομέα της ε, αστυνομικής συνεργασίας, δικαιοσύνης και πληροφοριών. Το κράτος δικαίου είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα πρέπει να έχει την προσοχή μας. Και σήμερα βλέπουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι το να είναι ανεξάρτητες οι δικαστικές αρχές όταν το σύστημα δηλαδή λειτουργεί. Τέλος, θα πρέπει να δούμε και τις εξωτερικές σχέσεις, το τομέα της δικαιοσύνης, ασφάλειας και δικαιοσύνη και στις εξωτερικές σχέσεις, διατλαντικές σχέσεις πιο συγκεκριμένα και σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες. Και άλλο ένα θέμα που δεν είναι θέμα πολιτικής μα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς υιοθετούμε μέτρα πολιτικής, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μας με μεγάλη επιμέλεια και πέφτουν όλα μέσα σε ένα μαύρο κουτί στο Συμβούλιο και κολλάνε εκεί. Υπάρχουν μέτρα που δέκα χρόνια τώρα έχουν κολλήσει για τη διαφάνεια, οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης, πολιτικές για το άσυλο. Είναι απαράδεκτο να κολλάνε όλα στο Συμβούλιο. Προσπαθούμε να αντισταθμίζουμε για αυτά τα οποία δεν προχωράνε, υιοθετώντα νέε πολιτικέ, ενώ πρέπει είναι προτιμότερο να εστιάσουμε την προσοχή μας στις πολιτικές ε, οι οποίες ε, εγκρίνονται, ώστε να περάσουν από το Συμβούλιο και να υλοποιούνται στα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε κυρία Ιντουέλ, κυρία Ρέντκε. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά σημαντικά σημεία ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι. Η Επιτροπή μας νομίζω ότι βρίσκεται στο προσκήνιο των πολύ σημαντικών συζητήσεων που θα ακολουθήσουν στη θητεία αυτή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο ευρύτατο χαρτοφυλάκιό μας, στα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Συμφωνώ ότι είδαμε στο παρελθόν ότι αν δεν σπρώξει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο πολύ συχνά μας μπλοκάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει. Αλλά για τα θέματα που μας απασχολούν πρέπει να παραγάγει αποτελέσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το περιμένουν οι πολίτες. Προσπάθησα να βάλω σε μια σειρά τις σκέψεις τις οποίες αναφέραμε στην πολιτική μας ομάδα για τις προτεραιότητες της ομάδας και νομίζω καταρχήν θέλουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό θα έχει κεντρική σημασία. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ελέγχου και αξιολόγησης του κράτους δικαίου και αν υπάρχουν παραβιάσεις να λαμβάνονται μέτρα να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του άρθρου 7 και της διαδικασίας την οποία έχει επιδιώξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, οδηγία που έχει προωθεί από το Κοινοβούλιο κατά της βίας, κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν πολλοί ακτιβιστές οι οποίοι περιμένουν από την Επιτροπή μας ε, να κάνουμε κάτι για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά τους. Ένα σύστημα ασύλου είναι το επόμενο θέμα με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ τονίζω το πόσο ανησυχούν οι συνάδελφοι για το πακέτο για τη δέσμη μέτρων για το άσυλο. Πιστεύω ότι παλέψαμε πολύ στην προηγούμενη θητεία για να βρεθεί μια συμβαστική λύση μεταξύ του φάσματος των πολιτικών ομάδων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και δεν μπορεί να παραμείνει αυτό κρυμμένο στο Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Έρευνα και διάσωση, και αυτό είναι μια προτεραιότητα, και η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης γιατί δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε σε συμφωνίες για τη μετανάστευση ε, να υπονομεύουν το δικαίωμα ε, εξέτασης που έχει το δικό μας κοινοβούλιο. Επίσης, η προάσπιση της ασφάλειας χωρίς να ξεχνάμε τα πολιτικά δικαιώματα και λαμβάνοντα υπόψη και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα θέματα αυτά. Βλέποντας και τις ακροάσεις με τους νέους επιτρόπους, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για το 1 τέταρτο της νομοθεσίας σε αυτό το Κοινοβούλιο. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για ε, τους τίτλους των χαρτοφυλακίων και πρέπει να φροντίσουμε ότι κατά τις ακροάσεις θα έχουμε πολύ προσεκτικό έλεγχο των αρμοδιοτήτων. Να κοιτάξουμε πέρα από τις λέξεις και τους τίτλους ε, το πραγματικό αντικείμενο των πολιτικών που πρόκειται να, ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ρένκε. Εκ μέρους της ID. Δεν είναι εδώ η κυρία Ταρντίνο. Α, εσείς. Συνάδελφοι. E θα μιλήσω συνήθω στην ε, Μητρική μου γλώσσα. Νομίζω όταν μιλάμε για χάραξη πολιτικών θα πρέπει να εξετάζουμε σε τι συγκυρία βρισκόμαστε εμεί οι βουλευτέ. Και σύμφωνα με τον ε, ΟΗΕ, ε, από ένα θα πάει στα τέσσερα δις ο πληθυσμό της Αφρικής και οι εθνογράφοι λένε ότι πάνω από τους μισούς Αφρικανούς είναι κάτω από 25 ετών και θέλουν να καταλήψουν την Ήπειρο Πού θα πάνε στην Ευρώπη. Επομένως εδώ έχουμε ένα διπλό δράμα, διότι χάνει ελληνικά χέρια, χάνει τη μεσαία τάξη η Αφρική, ε, στερείται οικονομική ανάπτυξη, έτσι ε, στερείται την ευημερία, όλος ο πληθυσμός. Ε, όμως, επίσης, έχουμε έτσι και εντάσεις πολιτιστικές στην Ευρώπη. Ε, οπότε, Αντί να έχουμε τον εμπλουτισμό, τον ε, πολιτιστικό, ε, έχουμε ε, μια αντιπαράθεση, έναν διαχωρισμό, αυτό που λέμε για το Ισλάμ. Επομένως, ποιος ωφελείται από όλα αυτά, τι προβλήματα λύνονται με το να ανοίγουμε διάπλατα τις πύλες. Το θέμα είναι επομένως η ασφάλεια. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωής μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε στο σπίτι μας μία μειονότητα. Θα πρέπει να μπει φρένο στη μετανάστευση, να η πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό όχι επειδή θέλουμε να είμαστε σκληροί προς τους μετανάστες, αλλά το λέω αυτό από αγάπη για τους δικούς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε και πάμε τώρα για το ECR στον κύριο Προκατσίνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας ομολογώ ακόμα. Δεν έχω αρκετή κοινοβουλευτική πείρα για να μπορέσω να συμβάλλω στην μεθοδολογία που θα χαράξουμε για να είναι όσο πιο αποτελεσματική η δραστηριότητά μας. Καλά πήγα και στο τελευταία συνάντηση των ε, ε, συντονιστών και από εκεί δανείζομαι ε, ό,τι εμπειρία μπορώ. Πάντως θέλω να πω ότι αυτή η Επιτροπή είναι σίγουρο ότι είναι αυτή που έχει την πιο μεγάλη πολυφωνία. Όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις ακριβώς γιατί είναι τα πιο πολυσυζητημένα θέματα αυτά που συζητούμε και το περισσότερο πολυσυζητημένο είναι η μετανάστευση. Επομένως, το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να τύχει ε, διαχείρισης. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να φερόμαστε κατασταλτικά και ότι είναι δυνατόν να φρενάρουμε την λάθρομετανάστευση για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Μα την νόμιμη μετανάστευση τη χρειαζόμαστε, όπως όλα τα κράτη τη χρειάζονται. Επομένως, αυτό πρέπει να κάνουμε, να φρενάρουμε την παράνομη μετανάστευση και να προστατεύσουμε αυτούς που φεύγουν για να γλιτώσουν από διώξεις και από πολέμους, να μην τους αφήνουμε στην τύχη τους τι πρεσβεύουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα διαφορετικό προβλέψιμο, όπως λένε, σύστημα ασύλου. Ο επαναπατρισμός των λαθρομεταναστών ε, πρέπει να γίνει μέσω μιας διαφορετικής ε, προσέγγισης. Όχι, όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καλούς και κακούς. Σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ποιος έχει διαφορετική άποψη, ποιος έχει διαφορετικά και τι πρέπει να γίνει για όλους. Άλλες προτεραιότητες, ξέρετε ότι έχουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα και όσον αφορά την ασφάλεια θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το ριζοσπαστισμό όχι μόνο με πολιτική ασφάλειας αλλά και με πολιτιστικά μέσα με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και τελικά θα πρέπει να προωθηθεί η πρόταση Λέναρτς ούτω ώστε να θωρακίσουμε τις ε, βάσει δεδομένων ε, της ε, Eurodac. Έχουμε πολυφωνία εδώ, διαφορετικές απόψεις, αλλά όσο και αυτό φαίνεται αυτονόητο, νομίζω τελικά θέλουμε όλοι το ίδιο. Η κυρία Ένστ για την ΚΟΥΕ. Να ζητήσω συγγνώμη που άργησα, όμως ε, υπήρχαν πραγματικοί λόγοι που με οδήγησαν στην καθυστέρηση. Τώρα, για τις προτεραιότητες ε, που θα θέλαμε εμείς να καθοριστούν και που για μας είναι πολύ σημαντικές, φυσικά το πρώτο, η πρώτη προτεραιότητα για μας είναι το άσυλο και η μετανάστευση. Κάτι που ακόμη μας λείπει και που πρέπει να το συζητήσουμε και, και νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Το ερώτημα είναι μπορούμε να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε την νόμιμη μετανάσταση. Ποια μέτρα θα μπορούσαμε να λάβουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια συστήματα πρέπει να αναπτύξουμε για να εξυπηρετηθεί ένα τέτοιο στόχο και πώ μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό με έναν τρόπο μη γραφειοκρατικό. Και μετά βεβαίω υπάρχει η, θεματική του ασύλου. Κάποια ε, κράτη-μέλη έχουν ήδη ε, συνάψει μια συμφωνία για την ε, καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες ε, για τη διάσωση και την ανέβρεση ώστε να εντοπίζεται για παράδειγμα κάποιο πλοιάριο στα ανοιχτά της Μεσογείου, στα ανοιχτά της Λιβύης και να το επιστρέφει, να επιστρέφει στη Λιβύη. Και πώς στην πράξη τελικά θα εξασφαλίζεται το δικαίωμα των ε, ανθρώπων να υποβάλουν αίτημα ε, χορήγησης ασύλου, πώς μπορεί να έχουν ε, καλές πιθανότητες να λάβουν άσυλο. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν τα έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση αντιπαραθετική με τον κανονισμό του Δουβλίνου, Υπάρχει μια καλή πρόταση που βγήκε από εδώ μέσα από το Κοινοβούλιο ε, και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν ε, ασχολείται με την πρόταση αυτή του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο με τη σοβαρότητα που ε, του αρμόζει. Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται συνεργασία όλων των κρατών μελών. Μετά, παρακολουθήσεις, μαζική παρακολούθηση των πολιτών. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα ε, που μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο και που θεωρούμε ότι ενισχύεται γιατί ακριβώς συνδέεται και με το ζήτημα, των, ε, ε, με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επίσης νομίζουμε ότι είναι αποφασιστική σημασία. Νομίζω ότι μπορούμε σε διάφορα θέματα, σε διάφορους φακέλους να διαπιστώσει κανείς ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία σε αυτή τη θεματική, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλύψαμε το έδαφος για τους ε, συντονιστές. Ήδη ε, προλέγει το έδαφος, η προηγούμενη συζήτηση, οι συζητήσεις και η συζήτηση των συντονιστών που θα τα πούνε και αύριο. Αλλά τώρα ε, ήρθε η ώρα της γενικής συζήτησης που ακριβώς αυτό ήταν το νόημα αυτού του σημείου σήμερα σε διάταξη. Όποιο θέλει μπορεί να λάβει το λόγο από τους συναδέλφους. Από ό,τι βλέπω ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι. Οπότε ε, ε έχουν διάφορες Και στο λόγο, ε, με τη σειρά θα λάβει το λόγο, Στάτνερ. Ευχαριστώ. Να σημειώσω καταρχάς ότι η συζήτηση για τις προτεραιότητες για μας και για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αφενός Αποδεικνύει η συζήτηση αυτή ότι επιλέγουμε δημοκρατική προσέγγιση και ότι συζητάμε πραγματικά ποιε είναι οι προτεραιότητε μα. Επίση, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων είναι μια επιτροπή με πολύ ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων. Ουσιώδη όμω είναι τα θέματα που συζητάμε όχι μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά για την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί αυτά που αποφασίζονται εδώ έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων ασχολούμαστε μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι, η ασφάλεια, η ασφάλεια. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει και ελευθερία. Και αυτό το βλέπουμε και στη συζήτηση που έγινε για τους ε, ε, ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Φυσικά ε, δεν θέλουμε κανένας μας να γίνονται έλεγχοι συνοριακοί στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θέλουμε μια ελεύθερη αγορά, ελεύθερη κινητικότητα ε, αλλά για να μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει στην πράξη χρειάζεται καλή προστασία των εξωτερικών συνόρων και μετά τη μεταναστευτική κρίση 2015-2016 διαπιστώσαμε όλοι μας ότι η ασφάλεια είναι πραγματικά προϋπόθεση για την ελευθερία. Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση και οι πολίτες περιμένουν από εμάς να δώσουμε επιτέλους σοβαρές απαντήσεις σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Εδώ λοιπόν θα κληθούμε να ασκήσουμε πίεση στην Επιτροπή Φοντερ Λάιεν ακριβώς για να οδηγηθούμε στην ενίσχυση του προσωπικού και του προϋπολογισμού της Frontex με 10.000 άτομα συγκεκριμένα και για να κλείσουν επιτέλους τα κενά ανάμεσα στη χορήγηση ασύλου και στις επιστροφές. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις που έγιναν χθε στην ε, Μάλτα αποδεικνύουν ότι τα όσα έχουν γίνει αυτή τη στιγμή δεν αρκούν, δεν εμποδίζουν τους διακινητές, αντιθέτως τους ε, ρίχνουν νερό στο μήλο των διακινητών οι στάσεις των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης της ίδιας. Τέλος, προστασία προσωπικών δεδομένων και κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Κυβερνοεπιθέσεις δεν θα γίνονται πια μόνο στις ταινίε επιστημονική φαντασία, αλλά και στην καθημερινότητά μα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε καλύτερε υποδομέ για καλύτερη προστασία των πολιτών. Και επίση ζητούμενο ε, είναι να συζητηθεί και το θέμα της, ε, του κράτους δικαίου που είναι ένα από τα βασικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι βασιζόμαστε στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος, το κράτος δικαίου. Κάθε προσπάθεια υπαναχώρησης, οπισθοδρόμησης πρέπει να ανακοπεί. Πρέπει να είμαστε και μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το κράτος δικαίου και στο εσωτερικό και προς το εξωτερικό. Και τέλος, η όλο ένα και μεγαλύτερη απειλή της τρομοκρατίας που προσπαθεί να αξιοποιήσει τα παραθυράκια και τα κενά που υπάρχουν και στην Ευρώπη. Και εδώ χρειάζεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπόλ θα έχει τα φόντα και τα μέσα για να μας προστατεύει. Ακριβώς για να εξασφαλίζει τις, αυτά που θέλουμε όλοι μας. Ασφάλεια και ελευθερία. Ευχαριστώ κύριε Στάτλερ Κυρία Πούντεκ, η σειρά σας. Παρακαλώ. Ε, δύο λεπτάκια αν μπορείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα κάνω που είπατε. Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά είναι η κύριε προτεραιότητα. Τελικά, αυτά είναι το πλαίσιο στο σώμα δικαίου για το οποίο και συζητούμε. Αλλά αυτό θα πρέπει να κάνουμε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, για μια περιοχή ε, ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. Ε, θα πρέπει να δούμε το ότι όλο ένα και περισσότερο επί των δικαιωμάτων ασκεί επιρροή αυτή η πολιτική, αυτές οι πολιτικές. Ήμουν διαμεσολαβητήρα στην Πολωνία, οπότε θέλω να υπάρχει ισότητα για όλους όσον αφορά τα δικαιώματα και θα πρέπει να δούμε τώρα τι μέσα πολιτικής θα έχουμε, οπότε ε, γι' αυτό σας λέω να εστιαστούμε στα δικαιώματα ε, των ανθρώπων. Μια αναπηρία, ισότητα ε, των δύο φίλων, βία των γυναικών, μετανάστερα. Αυτοί, αυτές είναι οι βάλλοντας πολιτικές ομάδες και δεν είναι θωρακισμένες όσον αφορά τη δυσμενή διάκριση γιατί πολλές φορές τα δικαστήρια δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα και δεν υπάρχει διαίρεση των εξουσιών. Οπότε θα πρέπει να δούμε ε, το ότι χρειάζεται να εξαρτήσουμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με το κράτος δικαίου. Γιατί μόνο μόνο οι ποινές ε, δουλεύουν κατά των λαϊκιστών. Αλλά, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να πλήσουν ε, τον κοσμάκι γιατί δεν φταίει αυτός. Κύριε Αλτσαλάνη. Κυρία, κυρία, συμπαθάτε με. Κύριε Λτσαλάνη. Δεν πειράζει, πρόεδρε, δεν πειράζει να σας τα πω στα σουηδικά. Ε, ευχαριστώ έτσι για ψυχαγωγία. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ε, αναφέρθηκαν ήδη πάρα πολύ σημαντικέ ε, πολιτικές ε, και συμφωνώ 100% ευχαρίστω. αλλά υπάρχει κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πολύ και αυτό είναι η καταπολέμηση ε, πάσης φύσεως ρατσισμού. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι είμαστε δημοκρατική κοινωνία εάν οι πολίτες μας δεν χαιρούν ισότητα και όλα εξαρτώνται από το χρώμα του δέρματος και από αυτό εξαρτάται το αν θα βρουν δουλειά, ε, το τι μεταχείριση θα έχουν αντισημιτισμός, ε, ισλαμοφοβία, αφροφοβία όλα αυτά θα πρέπει να θεωρήσουμε την πρωτεύουσα της Επιτροπής μας κυρία Τικ. Ευχαριστώ πρόεδρε, Η κυρία Στρίκ. Περιλημμένα, είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την καινούργια συμφωνία για το πλαίσιο. Κύριε Φόντερ Λάιεν, ήδη τα έχει εξαγγείλει όλα αυτά. Γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε μεγάλη απογοήτευση διότι τα κράτη-μέλη, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το περιεχόμενο. Και επιμένω. Ω ΛΥΜΠΕ, θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τη πρώτα-πρώτα, να κάνει κάποια μελέτη του κατά πόσο εφαρμόζεται η ισχύουσα πολιτική για το άσυλο και Περιμένουμε τώρα, ήδη εδώ και πολύ καιρό, για τέσσερι εκθέσει εφαρμογή για τέσσερα μέσα πολιτική ασύλου. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουν προ αυτή την κατεύθυνση. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε κάποιε πολιτικέ που στοιχεία ε, και θα έρθει η ώρα για τούτο όταν θα πρέπει να συμβάλλουμε σε μια συμφωνία. Τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι δυσκολεύονται να συναντήσουν όσον αφορά την εσωτερική διάσταση και ε, συμφωνούν για την εξωτερική διάσταση του θέματος, συμφωνούν για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, για το πώς θα σταματήσουν τους μετανάστες να μην ε, έρχονται, να μην υπάρχει επανεισδοχή, αλλά ε, το, κάνω αυτό και για πρόσφυγες που είναι ανεγνωρισμένο ότι χρειάζονται προστασία και συμφωνούν για το πώς θα πάνε σε τρίτες χώρε Να, Εξού και συμφωνία με την Τουρκία. Άρα είναι μια βαριά ευθύνη αυτή. Και τι κάνουμε, τη μεταθέτουμε σε τρίτες χώρες. Νομίζω ότι η ΛΥΜΠΕ έχει πολλά επιχειρήματα για να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε προσεκτικά αυτή την πολιτική. Δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης σε επίπεδο παγκόσμιο. Είναι θέμα προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν έχουν όλε οι χώρε σύστημα ασύλου. Γιατί αυτό χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μια βιώσιμη, μια διαρκή προστασία. Σε πολλές χώρες ε, ε, είναι αμφίβολο το αν υπάρχει κράτος δικαίου γιατί υπάρχει διαφθορά, άρα θα πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά έχουν σοβαρές συνέπειες για τους συνέπειες. Ό,τι συμφωνήσουμε θα έχει επιπτώσεις στην τύχη, όπως και συμφωνείς με τις τρίτες χώρες. Είναι επίσης θέμα θεσμική Είναι παράδοξο το Κοινοβούλιο να μην παίζει ένα σημαντικό ρόλο παρά το ότι είμαστε αρχή του προπολογισμού. Ε, όμως, όμως, ο προϋπολογισμός είναι στην αρμοδιότητα όλων των ε, επιτροπών. Άρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι γίνεται με την εξωτερική πλευρά της ε, μεταναστευτικής πολιτικής. Ελπίζω αυτό ε, τώρα για τη θητεία τούτη θα γίνει προτεραιότητά μας. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται πλευράς νομικής, τι θα γίνει με τα εργασιακά θέματα για τους νόμιμους μετανάστες. Αυτό είναι δημοκρατική πρόοδος, δημοκρατική εξέλιξη. Θα είναι πιο λογική η εργασιακή πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση. Και ε, αυτό ωφελεί και το θέμα του ασύλου, αλλά όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Εκτός μικροφώνου. Ο πρόεδρος δεν ακούγεται. Δίνει το λόγο στον επόμενο. Κύριος Ούρικο. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώσαμε μια ενδιαφέρουσα έκθεση κατά του ρατσισμού. Και όμως διαπιστώνω ότι οι μας δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κατά πολέμηση του ρατσισμού. Όμω, ο περισσότερο κόσμο υφίσταται δυσμενή διακρίσει. σω εσεί δεν το αισθάνεστε στο πετσί σα, αλλά αυτό σημαίνει να, στη Σλοβακία. Είχαμε κάποια προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο στόχος ήταν κάποιοι δήμοι και κοινότητες με πολλούς Ρωμά. Όμως τι γίνεται, τον 20ο αιώνα χρηματοδοτούμε κάποια χωριά επί τη βάση του χρώματος, του δέρματος, του πληθυσμού. Μα τι να πω στους συμπολίτες μου που δεν παίρνουν δεκάρα. Να τους πω ότι όλα τα λεφτά πάνε στους Ρωμά. Υπάρχει και στην κυβέρνηση κάποιος που ασχολείται μόνο με τα προγράμματα για τους Ρωμά. Στέγαση δωρεάν. Μα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι γίνεται με, τον υπόλοιπο, με την πλειονότητα του πληθυσμού. Μα στο τέλος θα μας κυνηγήσουν. Και έχουμε και ένα σωρό εγκλήματα που διαπράττουν η Ρωμά. Αλλά και να στραβαμάτει η αστυνομία γιατί φοβάται. Φοβάται να μην χαρακτηριστεί ρατσιστική. Ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία ανακοίνωσε επισήμως ότι οι απειλές είναι κομμάτι του πολιτισμού των τσιγκάνων. Η απειλή κατά τη ζωής των άλλων. Μα πώς να ζήσει κανείς έτσι σε τέτοια χωριά. Να επιτίθενται στα παιδιά μας. Μόνο και μόνο γιατί δεν είναι τσιγκανάκια. Θέλω αντικειμενικότητα. Αυτό είναι φάρσα, δεν είναι αντιρατζιστική πολιτική που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν πειράζει ένα κομμάτι του πληθυσμού και όλοι οι άλλοι θεωρούνται ένοχοι. Ε, όχι, ας κάνουμε αντιρατζιστική πολιτική αντικειμενικά, αλλιώς το πράγμα θα γιάσει μη κατάληξη. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι ζητούν το λόγο. Πρέπει να σας πω ότι μετά την παρατήρησή σας, να σας πω ότι και εγώ ε, που είμαι από την Ισπανία, ε, Υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που είναι Ρώμα που δεν αποτελούν καθόλου απειλή για μας και για την ταυτότητά μας. Κατά κανένα τρόπο δεν αποτελούν απειλή οι Ρώμα. Ο κύριος Σανσαλέχος έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτως με αυτό το οποίο μόλις είπατε. Όταν σκεφτόμαστε το μέλλον, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι αυτό το οποίο εξελίσσεται τη στιγμή που κάνουμε σχέδια για το μέλλον και θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε σε απρόβλεπτες συνθήκες που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Τα επόμενα χρόνια η ψηφιοποίηση συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και για την εγκληματική δραστηριότητα. Δηλαδή, οι εγκληματίες όχι μόνο θα δραστηριοποιούνται σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά θα αλλάξουν και οι δικές τους δραστηριότητες θα προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, χρειαζόμαστε καλύτερη υλοποίηση και εκτέλεση αποφάσεων. Και αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαίνει συνεργασία. Και για τη συνεργασία χρειάζεται εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και οπωσδήποτε το ένταλμα σύλληψης, αν βελτιωθεί, αποτελεί μια πρόοδο, αλλά θα πρέπει και αλλού να προχωρήσουμε και άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους, ούτως ώστε να συσφίξουμε τις ε, σχέσεις μας ε, με τα Εθνικά Κοινοβουλία, εμείς ως ΛΥΜΠΕ. Και έτσι να εξαντλήσουμε τα περιθώρια που υπάρχουν για να κάνουμε βήματα προόδου. Μορένο, Σάντσες, έχετε το λόγο. Όχι, δεν ζήτησα το λόγο, πρόεδρε, αλλά δεν πειράζει. Απ. Α, όχι, δεν γίνεται. Ε, σας είχαν σήμερα, τέλος πάντων. Ευχαρίστω να σας τα πω για τις πατριότητες. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε και ο προλαλής σας και ο λέγω. Και βέβαια να σας πω τηλεγραφικά για τις προτεραιότητες, θα πρέπει να βάλουμε την μετανάστευση στις θα πρέπει να σταματήσει να είναι νεκροταφείο ή Μεσόγειος και επίσης ας εστιαστούμε σε κάτι που είναι ντροπή για την Ευρώπη. Τότε χιλιάδες νέων και παιδιών μένουν χωρίς μέλλον εδώ στην Ευρώπη. Αυτό που λέμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους ασυνόδευτους θα πρέπει αυτά εδώ τα παιδιά να μην βρίσκονται σε κάποιο κενό δικαίου. Και ε, επίσης στην περασμένη θητεία κάναμε πολλή δουλειά αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε, να μην επαναπαυθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε και για τον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Επίσης, να δούμε τι γίνεται το κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες και δεν εξαιρώ τη δική μου χώρα, την Ισπανία. Σεβασμός προς το κράτος δικαίου επίσης, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Λέμε ένα σωρό πράγματα τελευταία, αλλά είχα την ευκαιρία πριν εδώ που ήμουν πάλι στο Κοινοβούλιο να δουλέψω πάνω σε αυτό το ζήτημα και ακριβώς η προξενική προστασία είναι θέμα που ακόμα χρειάζεται ε, δουλειά. Αυτά τηλεγραφικά, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, για και δεν τον ζήτησα. Αλλά πάλι καλά, γιατί ήταν σημαντικό. Μα σα είχαν πιστέψει, μη ήσασταν σημειωμένο εδώ στη λίστα των αγορήτων. τέλο. Πάμε τώρα στον κύριο Αδάμοβιτσα. Κύριε Αντάμοβιτσα. Κυρία, κυρία. Και πάλι και εσείς με συγχωρείτε, λέει στην κυρία Ντάμοβιτ ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης για τις προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ κατά την επόμενη θητεία, Θέλω να αναφέρω ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Είναι η καταπολέμηση ε, των εκφράσεων μίσους και της ρητορικής μίσους. Θα έχετε προσέξει την κονκάρδα που φοράω με την ε, κόκκινη καρδιά. Είναι μια κονκάρδα κατά της ρητορικής του μίσους. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα. Αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεπαρκή. Η υφιστάμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η απόφαση πλαίσιο από το 2008 για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ε, δεν είναι επαρκής. Ορίζεται βέβαια η ρητορική του μίσους, αλλά περιορίζεται σε λίγα θέματα όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο επιθετικός εθνικισμός η εχθρική αντιμετώπιση των ξένων, αν το ερμηνεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο όμως, αφήνουμε απ' έξω ένα ευρύ φάσμα και προσώπων και φαινομένων. Η ρητορική του μίσους όμως επηρεάζει τους πάντες, όχι μόνο πολιτικοί αλλά και νέοι και ηλικιωμένοι και μαθητές του σχολείου, άτομα με αναπηρίες και άτομα χωρίς αναπηρίες, όλοι επηρεάζονται. Πρέπει να μιλάμε λοιπόν για απαλλαγή από την ρητορική του μίσους. Στο μέλλον θα πρέπει στην νομοθεσία μας να συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες που πλήττονται. Το Νοέμβριο η Επιτροπή μας προγραμματίζει μία δημόσια ακρόαση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, για την ελευθερία του λόγου, την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και στο διαδίκτυο και γενικότερα. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και μια ευκαιρία να θέσουμε φιλόδοξους στόχους ακριβώς για την καταπολέμηση της ρητορική του μίσους και στο διαδίκτυο και εκτός. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σε αυτή την ακρόαση να συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο και τις επιπτώσεις στην κοινωνία. Η παραπληροφόρηση, οι ψευδείς ειδήσει είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά και μπορεί να έχει πολύ επικίνδυνες συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να συστηθώ. Ε, μάλλον δεν χρειάζεται να σας συστηθώ. Ξέρετε ότι δουλεύω στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου πάνω από τρία χρόνια. Πρώτα ως ε, γιατρός και συνέχεια και ως ε, αξιωματούχος στη Λαμπεδούζα. Τώρα πια έχω την ευκαιρία και εργάζομαι επί της μεταρρύθμισης του κανονισμού του Δουβλίνου, του συστήματος του Δουβλίνου, συγγνώμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, να προχωρήσει για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα λειτουργικό σύστημα ασύλου. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο έγινε στη Σύνοδο Κορυφής της ε, Μάλτας πριν από λίγες μέρες. Ακριβώς γιατί επιχειρείται για πρώτη φορά να συγκροτηθούν κάποιες κοινέ δομές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με προσωρινά, προαιρετικά, εθελοντικά μέτρα. Όταν η κατάσταση είναι αυτή που είναι στη Μεσόγεια, Μεσόγειο χρειαζόμαστε εντοπισμό και διάσωση πανευρωπαϊκών διαστάσεων. Γιατί έχω δει ανθρώπους να πνίγονται, να πεθαίνουν, είδαν πάρα, είδα πολλά παιδιά και αυτό είναι, είναι μια κατάσταση τελείως απαράδεκτη, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν το μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να διασώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Έχουν ήδη πεθάνει 40.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο. Παιδιά σαν τα δικά μας. Και αυτό διότι δεν υπήρχε ένας μηχανισμός εντοπισμού και διάσωσης. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πεπισμένος ότι μία από τις προτεραιότητες μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ε, νόμιμων οδών μετανάστευσης. Και για εκείνους που ε, δικαιούνται διεθνή προστασία, αλλά και για τους οικονομικούς μετανάστες. Και δεν μιλάμε για υψηλά εξειδικευμένου μετανάστε μόνο. Μιλάμε για οικονομικού μετανάστε. Ναι, είναι οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα στι χώρε του. Έχουν και αυτοί δικαίωμα στη μετανάστευση. Είναι σημαντικό λοιπόν να προχωρήσουμε με την τροποποίηση της οδηγίας του 2002 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δημιουργούν τους δικούς τους τρόπους με τους οποίους βοηθούν τους αλληλείς τους, για παράδειγμα. Αυτό δεν πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να έχουν περιθώριο τα κράτη, να τα βοηθήσουμε να μπορέσουν να κάνουν κάτι για αυτούς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Άλλωστε, η Ευρώπη γεννήθηκε με θεμέλιο αυτές τις αρχές, τις αξίες, την φιλοξενία, την αλληλεγγύη. Αυτές είναι οι αξίες μας και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να βρούμε τις λύσεις. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπράγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα ακούστηκαν για τον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των όσων έχουν αποφασιστεί, αλλά και στην επιβολή του νόμου. Είναι σημαντικό ακριβώς για να δοθεί και μια αξιοπιστία σε όσα έχουν αποφασιστεί στο παρελθόν. Και νομίζω ότι επίσης πρέπει να χαράξουμε μια κόκκινη γραμμή για νέες προτάσεις ε, στον τομέα της ασφάλειας. Δεν θέλουμε μαζική παρακολούθηση ή συλλογή προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών. Όπως είναι η διατήρηση δεδομένων, PNR, SWIFTED γιατί αυτή η μαζική παρακολούθηση πραγματικά μεταφέρει το, τον συσχετισμό των δυνάμεων υπέρ των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσει είναι αυτέ που ελέγχουν του πολίτε αντί να συμβαίνει το αντίθετο. Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε μια δημοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μορατόριουμ για νέε προτάσει που θα αφορούν την ε, ασφάλεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ελευθερίες μας. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στη Νέα Επιτροπή, ότι ακριβώς αυτή την κόκκινη γραμμή περιμένουμε να την χαράξουν και εκείνοι και να τη σεβαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νέας θητείας. Ευχαριστώ, η κυρία Κάνκο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ε, αίσθημα που μου δημιουργείται όταν είμαι εδώ στη Λίμπε. σχεδόν ποτέ δεν ακούω τίποτα σχετικά με την ευθύνη που έχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είναι δική τους ευθύνη να, φροντί, να φροντίζουν τους, τον, λαό, τον, τον λαό τους. Εγώ όταν ήμουν παιδί ε, είχα όνειρο ο πρωθυπουργός της χώρας μου να κάνει τη δουλειά του. Υπήρχε μάλιστα ένας και τον σκοτώσανε. Οπότε, στο πλαίσιο αυτή της ευθύνη, της υπευθυνότητα, η κατάσταση είναι, είναι η εξή. Όταν μιλούμε για μεταναστευτική κρίση, δεν βλέπουμε τις χώρες προέλευση ως χώρες στι οποίε μπορούν να αναπτυχθούν. Και αυτό κανείς μπορεί να το ε, διαισθανθεί και στις πολιτικές που ακολουθούνται ε, στη Δύση. Δεν βλέπουμε τις χώρες αυτές ως αγορά, ως ε, χώρες με κάποιο δυναμικό. Γι αυτό, γιατί αν το κάναμε αυτό, θα είχαμε αρχίσει να ε, ακολουθούμε άλλες πολιτικές. Ξέρετε ότι στη δεκαετία του 70 ε, υπήρχαν μεγάλες ελπίδες για την Αφρική. Δυστυχώς δεν ευωδόθηκαν. Και τέλος, για τη μετανάστευση. Όταν ακούω κάποιους από εμά να μιλάμε για τους μετανάστες, ε, νιώθω ότι κάποια ε, μέρη του σώματός μου και του εγκεφάλι μου λείπουν. Ξέρετε, ήμουν και εγώ μετανάστρια. Έχουμε πολλές δυνατότητες και μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς στην κοινωνική ζωή. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλε αυτέ τι δυνατότητε που φέρνουν μαζί του οι μετανάστε. Γιατί φυσικά κάθε άνθρωπο έχει και ανάγκε, αλλά έχει και δυνατότητε να προσφέρει. Έτσι πρέπει να του τους δούμε του μετανάστε, έτσι θα καταφέρουμε να του εντάξουμε στι κοινωνίε μα. Και θέλω να τελειώσω λέγοντα ότι η ανησυχία μου είναι ότι όλοι μα θέλουμε λύσει. Έχουμε ενδεχομένω διαφορετικέ οπτικέ και διαφορετικέ ε, ιδέε. Όμω όλοι σε τελική ανάλυση θέλουμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση λύσεων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Ντελβοσκόρφιλντ. Oui. Euh, cela a déjà été évoqué par κυρία και χρειάζεται και η Λίμπε και το Κοινοβούλιο να προτάξει τις αρμοδιότητες του, τον ρόλο του να προβάλλει Μετά την εκθέση Αργεντίνη είδαμε τι έγινε όσον αφορά την πλειοψηφία μας ε, ότι το Συμβούλιο μας αγνόησε και άρα με την Φιλανδική Προεδρία είμαστε αποφασισμένοι αλλά δεν μας ακούνε, δεν μας λαμβάνουν υπόψη αυτό. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, σημαντικό προηγούμενο διότι η νομοθεσία που εδώ εγκρίνουμε αφού την επεξεργαζόμαστε ε, θα πρέπει να τη κάνει άλλη υποδοχή ε, στα πλαίσια όμως του αρθρού 7 είναι ακόμη περισσότερο σημαντικό εάν θέλουμε η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να είναι σοβαρή να παρέχει εγγυήσεις ε, δημοκρατίας, δικαιωμάτων, το κοινοβούλιο να έχει αρμοδιότητες που να γίνονται σεβαστές και ε, έτσι θα έχει μέλλον η Ευρώπη και το Κοινοβούλιο αν το Κοινοβούλιο λαμβάνεται υπόψη στα σοβαρά. Άρα θα πρέπει σε αυτή τη θητεία αυτά να κάνουμε, αυτά να προβάλλουμε, να μην έχουμε άλλες περιπτώσεις από την έκθεση της Αργεντίνη. Άρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο να κάνει τη φωνή του να ακούγεται. Σας ευχαριστώ. Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα του κράτους ε, δικαίου. Και δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες μας, πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ρόλο μας ως εποπτών, ως υπευθύνων για την επιτήρηση της κατάστασης του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το μέτρο με το οποίο θα κριθούμε δεν κρινόμαστε μόνο από το τι συζητάμε και τι ψηφίζουμε, αλλά και το τι τελικά εφαρμόζεται. Θα πρέπει να υπάρχει ενδελεχής έλεγχος όλων όσων αποφασίζουμε και ψηφίζουμε σχετικά με την εφαρμογή αυτών. Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή της νέας αυτής ε, πενταετούς θητείας και έχουμε όλο το χρόνο να το κάνουμε. Ξεκινάμε τη συζήτηση με ένα θέμα που αφορά τη μετανάστευση πολύ ε, σύντομα θα κατατηθεί και ένα νέο πακέτο το οποίο θα συζητήσουμε ενδελεχώς και σε βάθος. Θα πρέπει όμως ευθύ αμέσω να ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της εφαρμογής που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Μεσόγειο και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον τα πρόσφατα γεγονότα που είδαμε στην ε, Μεσόγεια, που πλέον ε, ε, είναι, βρίσκονται σαν κοιλίδες μαύρες στη συνείδηση και στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια του όταν πεθαίνουν άνθρωποι στην Μεσόγειο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ανοιχτό νεκροταφείο η Μεσόγειος και να κλείνουμε τα μάτια. Γι' αυτό και καλώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την σημασία που έχουν οι δραστηριότητες διάσωσης, να λάβουν σοβαρότατα υπόψη τους τη δουλειά που έχουν κάνει μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ακτιβιστές, τι έχει συμβεί με την ποινικοποίηση της παροχής βοήθειας και φροντίδας και υποστήριξης. Κάποιες φορές το πρόβλημα είναι η έλλειψη ανάληψης δράσης, η απουσία δράσης. Και νομίζω ότι και ο Πέτρο Μπαρτόλο είπε κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό, σε αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω και εγώ. Να δούμε την οδηγία του 2002. Και αυτό είναι το βασικό που θέλω να κρατήσετε από τη δική μου τοποθέτηση σήμερα. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουχαρέ, έχετε το λόγο. Deduzco, señor presidente, que, que soy yo. Μπουξαδέ. Μπουξαδέ, προφέρετε, πρόεδρε. Perdóname, perdona. Μπουξαδέ. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, eh, και σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς. Πάντα όταν μιλούμε για πρώτη φορά, ε, λέμε ότι για πρώτη φορά μιλάμε, καλά δεν μιλάω για πρώτη φορά, αλλά είμαι ε, καινούριο και ήρθα σε αυτή την Επιτροπή των Πολιτικών γιατί νομίζω ότι η ΛΥΜΠΕ είναι ακριβώς η Επιτροπή αυτή που ενσαρκώνει το αυθεντικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αυτό που το οποίο ιδρύθηκε, δηλαδή για τον ε, χώρο ε, δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας και επομένως είναι βέβαια θέματα τα οποία είναι φορτισμένα ιδεολογικά ε, που τα περιβάλλουν πάρα πολλές επιθέσεις, παραξηγήσεις και όλα αυτά αφορούν και, και καίνε όμω του πολίτε των κρατών μελών. Η ασφάλεια και η δικαιοσύνη εγγυώνται την ελευθερία των συμβολιτών μα αυτή που επίση είναι οι ψηφοφόροι μα. Επομένω. Ε, αυτά τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να αποτελέσουν τρόπο εγγυήσεων προς των δημοκρατικών ελευθεριών των ε, Ευρωπαίων ε, και να μπορούμε κάτι να κάνουμε για τους κινδύνους εις βάρος της ε, ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Άλλωστε, η ασφάλεια απειλείται άμεσα από τον εσωτερικό και διεθνή ε, ε, τρομοκράτη. Και ήδη είδατε τι έγινε στην Βαρκελόνη, ήδη έγινε κάποιο είδου σύλληψη ε, κάποιας συμμορίας τρομοκρατών με εννέα μέλη στην Βαρκελόνη. Οπότε θα πρέπει επίση να έχουμε εγγύσει για την δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πάει να πει η με θρησκευτική ευλάβεια εκτέλεση των ε, δικαστικών αποφάσεων. Και εγώ αυτό θέλω. Ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι αποφάσει και των αλλοδαπών δικαστηρίων. Τα αγγλικά δικαστήρια να αποφασίζουν να τα τηρούμε στην Ισπανία, επίση αν αποφασίζουν τα Ισπανικά να τα τηρούν όσα αποφασίζουν τα Ιταλικά ε, δικαστήρια, αλλιώ δεν έχει νόημα. Και οι ε, ψηφοφόροι μου, ε, βέβαια οι Ισπανοί είναι, αυτοί με εξέλιξαν και του χρόνου δεν είναι τα θέματα του ρατσισμού και της όντας των ε, φίλων. Εμείς από το 1978 έχουμε σύνταγμα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις περισσότερα κράτη όλων ημών που εγγυώνται αυτές τις ελευθερίες. Μα τι, τι, να, τι να κάνουμε παραπάνω. Όχι, μπορούμε όμως να εγγυηθούμε για τους ε, ε, συμπολίτε μας, να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου να μην ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Τώρα θέλω να πω για τους συναδέλφους, για όσα είπανε, αναφέρθηκαν για το ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε, θα πρέπει να έχουν πιο αποτελεσματικού μηχανισμούς ε, για αποφάσεων ε, για την Ευρωπαϊκή Αστυνομία και επίσης και για το νομοθέτημα για την Eurodac που έχουν αναλάβει τη σχετική έκθεση. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Έχει το λόγο τώρα ο Φέστ. Ευχαριστώ. Εγώ ήρθα σε αυτήν την επιτροπή με την ελπίδα να συζητάμε ζητήματα κράτου δικαίου, πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνη. Κάποιε φορέ όμω έχω την ε, αίσθηση ότι θα έπρεπε να, να μετονομαστεί η επιτροπή αυτή σε επιτροπή νόμιμη μετανάστευση και ασύλου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η μετανάστευση έρχεται όλο ένα και περισσότερο σε αντίθεση με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Εδώ αυξήθηκαν οι επιθέσεις εναντίον ομοφιλοφίλων, χριστιανών, εβραίων και γυναικών. Και αυτό είναι ε, κάτι που αποδεικνύεται και στατιστικά. Και αυτές οι επιθέσεις προέρχονται από μετανάστες, ιδίως από μουσουλμανικές χώρες. Οπότε έχουμε μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στη μετανάστευση και την προστασία των ε, πολιτικών ελευθεριών. Οπότε η Επιτροπή μας θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει ε, πει και η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιεν, δηλαδή την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ανοιχτή, ελεύθερη κοινωνία και αυτή δεν μπορεί να προστατευθεί ε, μέσω της ε, επινόησης ε, ένα και νέων ε, νόμιμων οδών μετανάστευσης αλλά με τη δημιουργία συγκεκριμένων διαδικασιών επιλογής και με το να πούμε κάποια στιγμή ότι όταν πια θα έχουμε γεμίσει θα κλείσουμε τα σύνορα. Αυτά πρέπει να είναι αυτά που θα μας ε, απασχολήσουν και ελπίζω αυτά να μην είναι μόνο τα θέματα που θα απασχολήσουν την Κομισιόν Φοντερ Λάιεν αλλά και τη δική μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σχιτβέγγι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Χαιρετίζω την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε αυτές τις προτεραιότητες ε, των εργασιών μας εδώ στο πλαίσιο της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής θητείας. Νομίζω ότι αυτή η συμπεριληπτική και συνεργατική μέθοδος προσέγγισης των θεμάτων θα είναι ε, η άγουσα που θα ακολουθήσουμε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Συζητάμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα και η ευθύνη που έχουμε είναι πάρα πολύ υψηλή. Γι' αυτό το να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο των προτεραιοτήτων ε, είναι βεβαίως σημαντικό, αλλά θέλω να πω και δύο ε, σκέψεις σχετικά με το πώς θα πρέπει μεθοδολογικά να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά κατά τη γνώμη μας στο έργο μας. Είναι σαφές ότι προφανώς εδώ σε αυτή την Επιτροπή συμμετέχουν άνθρωποι με πολύ διαφορετικές απόψεις, ιδίως σε θέματα όπως είναι αυτό της μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει κατά συνέπεια ότι σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορές μας και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει χώρος να εκφράζονται οι διαφορετικές απόψεις. Αυτή θα πρέπει νομίζω να είναι η αφετηρία όταν θα γίνονται οι συζητήσεις για θέματα όπως είναι η μετανάστευση και τα συναφή θέματα. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ε, ο ένας τρόπος ε, να εκφράσει κανείς την αλληλεγγύη του στους άλλους είναι η αποτελεσματική προστασία των ε, εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει κάνει η Ουγγαρία τα τελευταία λίγα χρόνια και κατά συνέπεια για μένα αυτό σημαίνει ότι συμβάλαμε και στην ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί και είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η ίδια προσέγγιση νομίζω ότι είναι απαραίτητη όταν συζητούμε του τρόπου παροχή βοήθεια. Κάποια στιγμή, ε, κάποιοι, ένας τρόπος μάλλον ε, είναι να αντιμετωπίσει, για να βοηθήσει κανείς, είναι να βοηθήσει εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη, να αναπτυχθούν προγράμματα στη Μεσή Ανατολή, στην Αφρική, με την οικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα τρόπο να δείξει κανεί την αλληλεγγύη του και ενδεχομένω είναι και καλύτερο τρόπο να δείχνει κανεί την αλληλεγγύη του την πραγματική από το να πει κανεί Ελάτε όλοι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι και πιο υπεύθυνο αυτό που προτείνω εγώ η ίδια μεθοδολογία νομίζω ότι ε, πρέπει να εφαρμόζεται και ε, όταν συζητούμε τα θέματα του κράτους δικαίου, που είναι μια κοινή αξία. Μόνο μέσω της στήρησης κοινών προτύπων και μέσω της αντικειμενικής προσέγγισης μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα όσον αφορά το κράτος δικαίου. Έτσι μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας και την πρόοδο συνολικά της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Θέλω να αναφέρω ορισμένου τομεί που ήδη αναφέρθηκαν, αλλά θέλω να επαναλάβω εφόσον συμφωνώ. Ένα από του τομεί που θεωρώ σημαντικό να συζητηθεί μέσα στην επόμενη θητεία είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με το κράτος δικαίου. Γιατί αν κοιτάξετε στην Ευρώπη, βλέπετε ότι εκεί που καταραίει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι ακριβώς εκεί όπου η ισχύς βρίσκεται στα χέρια των ακροδεξιών, λαϊκιστών δυνάμεων. Νομίζω κάποιο Σλοβάκο με από τη Σλοβακία, είπε ότι δεν είμαι ρατσιστή, αλλά... Και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν αρκεί να πούμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές. Το να πούμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές δεν μας κάνει και μη ρατσιστέ. Είναι το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους που κρίνει αν είμαστε ρατσιστές ή όχι. Το αν οι Ρωμά στη Σλοβακία δρούν κατά τον ΑΒ τρόπο, έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους με διαφορετική προέλευση. Αυτό μας κάνει ρατσιστές ή μη ρατσιστές. Και το να λέμε ότι άνθρωποι με κάποιο υπόβαθρο, με κάποιο κάποια φυλή ή ε, θρησκεία ε, έχουν κάποια συγκεκριμένη ε, ιδιότητα, αυτό μας κάνει ρατσιστές. Και θα ήθελα να πω ότι στη Σουηδία, από που προέρχομαι, η απειλή κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και της δημοκρατίας δεν είναι απειλή που προέρχεται από τους μετανάστες και πάλι είναι απειλή που προέρχεται από τα κόμματα της δεξιάς. Πριν από λίγες εβδομάδες στη Σουηδία, ένας δήμαρχος δεξιός αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν την σημαία με το ουράνιο τόξο οι κοινότητε των ΛΟΑΤΚ, Αυτό είναι μια απειλή κατά των δικαιωμάτων και κατά του κράτους δικαίου. Δεν είναι απειλή που προέρχεται από τους μετανάστες. Επίσης το θέμα της τρομοκρατίας, πολιτικής και θρησκευτικής τρομοκρατίας είναι το δεύτερο θέμα και το τρίτο η μετανάστευση. Δεν μπορεί όπως σήμερα κάποιες χώρες να αναλαμβάνουν τεράστιε ευθύνε και άλλες χώρες να λένε ότι δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη, αλλά θέλουμε να υποφελούμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη την οποία λαμβάνουμε κατά ποικίλου τρόπου. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας παράλληλα με την υποστήριξη την οποία λαμβάνουμε και καλώς ε, παρέχουμε ένα στον άλλον υποστήριξη ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια πραγματική ένωση και να μην καταρρεύσει όπως θα ήθελαν οι μη δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να θα μεν αφενός και να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας αφετέρου έναντι των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη γιατί και εγώ ίδια έχω υπόβαθρο μετανάστευση ε, και ειλικρινά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα αν οι γονεί μου και εγώ δεν είχαν υποχρεωθεί, εξαναγκαστεί να φύγουν από τη χώρα από την οποία προερχόμαστε. Δεν φεύγει κανεί από τη χώρα του γιατί θέλει να διασκεδάσει. Θα προτιμούσαν να μείνουν στη χώρα του οι μετανάστε, αλλά δεν μπορούν. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι εμεί απλώ αποφελούμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για αυτού που χρειάζονται βοήθεια. Έχετε καταλάβει διπλάσιο χρόνο μιλίες από αυτόν που δικαιούσε, λέει ο πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό και το πάθος σας, αλλά παρακαλώ συνοψίσετε. Τέλος, θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ασφαλής και νόμιμος τρόπος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην προσπαθούν ε, αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσουν παράνομους και μη ασφαλείς τρόπους. Άρα ασφαλής και νόμιμη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριος Μαγκίντ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια. Θέλω να πω ότι το 2008, πριν από πάνω από 11 χρόνια, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα οδηγία, την αποκαλούμενη οριζόντια οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης, για να εγγυηθεί την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ίσης μεταχείρισης, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά σε ευρύτατο φάσμα τομέων, ούτως ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση ε, με βάση τις πεπιθήσεις, τη θρησκεία ή τη φυλή. πρέπει να προωθήσουμε την ε, πρόοδο σε αυτούς τους τομείς, αλλά δυστυχώς αυτή η οδηγία παραμένει αδρανής. Η εκλεγήσα πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, δήλωσε ότι είναι πρόθυμη η νέα Επιτροπή να αναλάβει μέτρα και θα προτείνει μια νέα οδηγία κατά της διακριτικής μεταχείρισης που πρέπει και να αποτελέσει προτεραιότητα για την Επιτροπή μας. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να δώσει όθηση στο θεματολόγιο της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης και να εξασφαλίσει την προστασία κατά της διακριτικής μεταχείρισης σε όλους τους τομείς της ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο ο κύριος Στοντολάτσι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, για την ε, υλοποίηση που και η Σοφή το τόνισε στην αρχή. Πιστεύω ότι μία από τις προτεραιότητές μας πρέπει να είναι η ενίσχυση της δυνατότητας που έχει η Επιτροπή μας ε, να ασκεί τον έλεγχο της ε, εφαρμογής της νομοθεσίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τον Ιούνιο, όταν συζητούσαμε το πολιτικό πρόγραμμα που θα δώσουμε στον πρόεδρο της Επιτροπής, όλες οι ομάδες είχαν συμφωνήσει ότι ο έλεγχος ε, είναι μία από τις σημαντικές προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ε, πολιτικής του ασύλου και της μετανάστευσης και πρέπει να δούμε ε, τα σχετικά με την ε, υλοποίηση και της μέρημνας με βάση τις αποδείξεις. EBCJ θα πρέπει να είναι το evidence-based και θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα. Όταν μιλάμε για την ψηφιακή πολιτική, που είναι άλλη μια προτεραιότητα, πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η Επιτροπή μα, γιατί οι αρμοδιότητε για τον ψηφιακό τομέα καλύπτονται από πολλέ επιτροπέ. Δεν ανήκουν μόνο σε ένα χαρτοφυλάκιο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε καλή συνεργασία με τις άλλες επιτροπές που θα εξετάσουν την βιομηχανική πολιτική για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, για το 5G και εμείς στη Λίμπε να έχουμε σαφή πολιτική για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής πολιτικής. Το τρίτο σημείο είναι η εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης που ανεφαρθήκε από πολλούς συναδέλφους. Η ανησυχία μου έγκυται στο ότι θα έχουμε ένα επίτροπο για διεθνή συνεργασία στην ακρόαση του οποίου θα παίξουμε πολύ πολύ ίσονα ρόλο. Το μήνυμα το οποίο θα πρέπει ε, να περάσουμε είναι ότι μπορεί να έχουμε ίσονα ρόλο στην ακρόαση, αλλά ο έλεγχος τον οποίο θα ασκούμε θα είναι μείζονος σημασίας. Έχει πολύ σημασία για την Επιτροπή μας και θα πρέπει να δείξουμε με στεναρό τρόπο πόσο ε, κοντά θα είμαστε στην εκπλήρωση του καθήκοντός μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Φόλετ. Το πρώτο σημείο το οποίο ε, θέλω να πω είναι ότι ε, είμαστε 10 χρόνια δεσμευτικού χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει στην Επιτροπή μας να συζητήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και το πώς μπορούμε ε, να τα εξασφαλίζουμε ενεργά πολλοί ε, πλήττονται από τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, από περιορισμό της ελευθερίας του τύπου ε, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων και η συνεργασία τους με την κοινωνία των πολιτών είναι μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Μπορεί να κάνουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας για τον συρρυκνούμενο χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, παραδείγματος χάρη. Ένα δεύτερο σημείο, άσυλο και μετανάστευση. Και εδώ θα πρέπει επιγόντως ε, να τονίσουμε τη θέση την οποία ήδη έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ασκούμε συνεχώς πίεση στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό αλληλέγγυο σύστημα για το άσυλο και τη μετανάστευση. Και όταν λέω δίκαιο, θα, αυτό συμπεριλαμβάνει και την έννοια του ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για τη χορήγηση ασύλου χρειαζόμαστε επανεξέταση της οδηγίας για την διευκόλυνση, facilitation, γιατί υπάρχουν από τη μια μεριά οι άνθρωποι που ε, αναλαμβάνουν ευθύνη και προσπαθούν να ασχοληθούν με την έρευνα και διάσωση και από την άλλη πλευρά οι παράνομοι διακινητές και πρέπει να δούμε και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την βία και αντιμετωπίζουν στα δικά μας σύνορα βία και αρνητική αντιμετώπιση, εχθρική αντιμετώπιση. Χρειαζόμαστε ένα συνεχή έλεγχο των όσων γίνονται στα εξωτερικά σύνορα. Αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών μας σύνορων, αλλά παράλληλα χωρίς ε, να παραβιάζουμε τους δικούς μας νόμους, χωρίς να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητούμε τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και παράλληλα θα πρέπει να δείξουμε και εμείς την ίδια στάση στα εξωτερικά μας σύνορα και να μην παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν έχουμε νόμιμη οδό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Το ότι έκλεισε η οδός των Βαλκανίων ε, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα όπως οι ειδωμένοι ε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το δικαίωμα στο άσυλο και θα πρέπει να μεριμνήσουμε το δικαίωμα για το άσυλο να είναι πραγματικότητα όχι μόνο η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα, αλλά και η διαμονή των ετούντων άσυλο είναι ε, ένα από τα σοβαρά προβλήματα και πιστεύω ότι πρέπει να το θέσουμε ως θέμα. Και το θέμα του κράτους δικαίου είναι το επόμενο θέμα που θέλω να αναφέρω, παρότι το ανέφεραν και άλλοι ε, συνάδελφοι σήμερα, επειδή είναι σημαντικός ο ρόλος μας ε, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, πρέπει να το τονίσουμε. και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα για την αιρεσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ιδιαίτερα επικοδομητικής συζήτησης, που παρότι όταν ξεκίνησε η συνεδρίασή μας εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, δεν ε, είχαμε τόσες ελπίδες, τώρα θέλω να πω ότι ότι δύο συνάδελφοι που ήδη έχουν λάβει το λόγο ζήτησαν δευτερολογία, ζήτησαν ένα λεπτό παραπάνω. παρότι θέλουμε να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα σας δώσω το λόγο, αλλά να είστε πάρα πολύ σύντομοι, πιο σύντομοι από την πρώτη φορά. Μια και είναι η δευτερολογία σας αυτή τώρα. Κυρία Σίπελ και εσείς μετά. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ίσως υπήρξε κάποια παρανόηση κατά τη συζήτηση, έλαβα το λόγο και πάλι. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει χρήματα στους πρόσφυγες, στα χέρια τους δηλαδή, στους ίδιους τους πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά δίνουμε χρήματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν να βελτιώσουν την ένταξη διαφόρων ομάδων, μεταξύ των οποίων και η Ρωμά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ζητούν αυτή τη χρηματοδότηση και να υλοποιούν την ένταξη. Δεύτερον, δυστυχώς επειδή προέρχεται από τη δική μου χώρα, άκουσα κάποιες παρανοϊκές στατιστικές για το πόσο μη ασφαλέ είναι το να ζουν ε, στη Γερμανία οι γυναίκε ιδιαίτερα. Σα διαβεβαιώ ότι αισθάνομαι θαυμάσια και ελεύθερα να κυκλοφορώ στη χώρα μου και αυτέ οι στατιστικέ που ακούσαμε τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τι στατιστικές που διάβαζα εγώ οποτεδήποτε μέχρι τώρα. Τέλο, υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αναζητούν απασχόληση και θα ήταν καλό να μπορέσουν να βρουν δουλειά στι χώρε από τι οποίες προέρχονται, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους από τρίτες χώρες που θα δουλέψουν στις χώρες μας. Και σας λέω μάλιστα ότι ο Υπουργός Απασχόλησης της Γερμανίας έφτασε να πάει στο Μεξικό για να αναζητήσει εργαζομένους για την Γερμανία. Βεβαίως πολλοί φεύγουν από τις χώρες τους για να ξεφύγουν από, την, από τους διωγμούς και τα βασανιστήρια τι να τους πούμε, να μιλήσω στην κυβέρνησή σου μήπως και αλλάξει γνώμη και θελήσει τα επόμενα χρόνια να αλλάξει την πολιτική της. Όχι βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προστατεύσουμε, αλλά να μην ανακατεύουμε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κάποιο ζήτησε το λόγο πριν από τη δική σα δευτερολογία και μου ξέφυγε ο κύριος, ε, ε, και ο κύριος Βαντεντρίσε θέλει να δευτερολογήσει, αλλά ακούσουμε τον κύριο Βίντεκομ που ζήτησε το λόγο και μου διέφυγε. Κυρία Βίντεκομ, ζητώ συγγνώμη. Δεσποινής Βίντεκομ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε κάποιους δώσατε το λόγο δύο φορές και σε μένα ούτε μία πρώτη φορά. Και θέλω να πω ότι για πρώτη φορά λαμβάνω το λόγο στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι θα υπάρχουν αρκετές ε, ευκαιρίες, αλλά μόνο μέχρι το, την 31η Οκτωβρίου, γιατί μετά την 31η Οκτωβρίου ελπίζω ότι εγώ και οι συναδελφοί μου από το Ηνωμένο Βασίλειο θα λείπουμε, δεν θα είμαστε πια εδώ. Τώρα, μετά τη συζήτηση αυτή που ακούσαμε, θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές φοβίες και πολλές ωραίες λέξεις, αλλά αυτό το οποίο δεν συζητήσαμε είναι μια βασική απέτηση της δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε η ελεύθερη έκφραση, η ελευθερία του λόγου η ελευθερία του λόγου για οποιονδήποτε πολίτη, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό καθορίζει το αν μια δημοκρατία λειτουργεί ως δημοκρατία. Και μέσα στον ενθουσιασμό μας να προσπαθήσουμε να μην προσβάλλεται κανείς και να είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καταπατούμε την ελευθερία του λόγου. Και προσπαθούμε σχεδόν να ελέγξουμε και τη σκέψη γιατί μέσα από το λόγο προβάλλεται η σκέψη. Λυπούμε γιατί σε ολόκληρη αυτή τη συζήτηση δεν τονίστηκε το θέμα της ελευθερίας του λόγου. Βέβαια, τούτων λεχθέντων, νομίζω ότι δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περισσότερο θέμα του κάθε κράτους μέλους. Αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του να προστατεύσουμε αφενός τις απόψεις όλων, και αφετέρου να μπορούν όλοι να εκφράσουν τη γνώμη τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν από το κράτος τους. Ευχαριστώ κύριε Δεσποινής Βουίδεκο. Ο κύριος Βαντερντήσε. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, τα Ολλανδικά. Παρακολούθησα τη συζήτηση, τις τοποθετήσεις των ε, συναδέλφων και παρατήρησα κάποια πράγματα. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, ε παράδοξες ε, στάσεις. Εγώ το μόνο που έθεσα ως ερώτημα είναι ποιος ωφελείται από τη μαζική μετανάστευση. Πήρα μια απάντηση από το ΕΛΚ, από την ΚΟΕ, από τους φιλελεύθερους, από τους σοσιαλδημοκράτες και όλοι λένε ότι χρειαζόμαστε τους ανθρώπους αυτούς για να συνεχίσουν τα γρανάζια της οικονομίας μας να γυρνάνε. Μα πώς λειτουργεί η οικονομία. Μιλάμε για προσφορά και ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν ε, η προσφορά εργατικού δυναμικού μειώνεται, τότε αυξάνονται οι μισθοί. Όταν υπάρχει περισσότερη μετανάστευση, ασκείται πίεση στο ύψος των μισθών. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Και στη μετανάστευση, το θύμα της μετανάστευσης μάλλον είναι η μεσαία τάξη. Βεβαίως θαυμάσιο είναι να έχει κάνει μια ένωση με ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει τεράστια νεανική ανεργία ε, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και τι, τι ακούσαμε ότι κάνει η γερμανική κυβέρνηση φέρνει Μεξικανούς για να δουλέψουν. Και αυτό είναι κάτι που το υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό. Μετά, προστασία προσωπικών δεδομένων, πολιτικές ελευθερίες. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή και του λέει ότι ανοίγεται καινούργια θέματα ε, και προσθέτεται νέα στοιχεία στη συζήτηση. Παρακαλώ, αφού ζητήσατε δευτερολογία, φροντίστε να ε, συνεισφέρετε νέα στοιχεία, αυτά που δεν είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση. Ωραία, συνεχίζει ο Ελευθερία και ασφάλεια. Όσο περισσότεροι έλεγχοι διενεργούνται από τις κρατικές αρχές, τόσο καλύτερα. Είναι προϋπόθεση βεβαίως το να υπάρχουν έλεγχοι, ε, διότι όπως καταλαβαίνετε η μετανάστευση σημαίνει ετερογένεια. Άρα ε, υπάρχουν πολύπλοκα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύονται με την ενίσχυση των ελέγχων. Και εδώ έχουμε ακόμη και πρόβλημα ορισμών. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ωφελείται από τις πολιτικές μας η μία ή η άλλη ε, πληθυσμιακή ομάδα ή εθνοτική ομάδα. Γι' αυτό και θα πρέπει να επιμείνουμε στην εξέβρεση πολιτικών λύσεων τις οποίες μπορούν να αποδεχτούν όλες οι πλευρές. Εγώ ξαναλέω ότι μιλώ για τους παράνομους μετανάστες. Πρέπει να επιστρέφονται όλοι οι παράνομοι μετανάστες που έχουν έρθει στην Ευρώπη από την ε, Αφρική. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι το στίχημα που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να ε, ε, αναλάβουμε. Πρόεδρος, μου ζητήσατε δευτερολογία, παρακαλώ πολύ σύντομα όμως, γιατί ήδη συζητάμε εδώ και δύο, ε, ώρες. Παρακαλώ, κάντε μια δευτερολογία και θα προσπαθήσω εγώ να καταλήξω, να κάνω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Έχω να κάνω μια μικρή παρατήρηση στα όσα ακούστηκαν. Υπόθηκε ότι όταν άνθρωποι αντιμετωπίζουν ανάγκη, τότε θα πρέπει να γίνεται διαπραγμάτευση πρώτα και κύρια με τις κυβερνήσεις τους. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Μιλώ ως Ευρωβουλευτής και ως άτομο που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε φτωχή χώρα και έχω ζήσει πόσες και ποιες ελπίδες έχουν οι νέοι άνθρωποι. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους ε, στο, ε, στις στοχές χώρες, τους νέους ανθρώπους, τι περιμένετε από την Ευρώπη, τότε η απάντηση που παίρνει κανείς είναι γιατί ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίζει δικτατορίες. Φυσικά και πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε... που έχουν ανάγκη, που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποτρέψουμε, πώς θα εμποδίσουμε στο μέλλον ε, τη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων επικίνδυνων. Ίσως λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα καλύτερης ε, αξιοποίησης των μέσων που ήδη διαθέτουμε στην ε, οικονομική συνεργασία, στην, στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη, στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και στη διάσωση των ανθρώπων στη Μεσόγειο. Οπότε αυτό που πρέπει εμείς πάντοτε να εξασφαλίζουμε είναι ότι η δική μας προσέγγιση πραγματικά βοηθάει γόνιμα και επικοδομητικά στην επίλυση των προβλημάτων. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Τελικά φάνηκε ότι είχε νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τελικά υπήρχε, υπήρχαν πολλά θέματα που κάλυψαν μια σειρά από ε, ζητήματα και εκφράστηκαν, τοποθετήθηκαν ανοιχτά και δημοκρατικά όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Συζήτηση που θα τροφοδοτήσει και ε, θα, εμπλουτίσει και τη συζήτηση που θα γίνει στις ερυδρές των συντονιστών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και για την προετοιμασία των ακροώσεων των οριστέντων επιτρόπων. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω, σε σχέση με τη γενική προσέγγιση την οποία συζητήσαμε εδώ σήμερα, ότι δεν μπορώ να παρά να συμφωνήσω με τις απόψεις που, ε, εξέφρασαν κάποια από εσάς διαμαρτυρώμενοι σχετικά με το οργανωτικό σχήμα μέσω του οποίου προσεγγίζουμε τους ε, οριστέντες επιτρόπους που είναι και άμεσο αποτέλεσμα της, ε, του σχεδιασμού των νέων της νέας επιτροπής. Ε, σχεδιασμός που ε, βαρύνει την ε, εκλεγήσα πρόεδρο, την κυρία Φόντερ Λάιεν. Κύριε Τουντοράση, το είπατε ότι και έχετε δίκιο ότι κάποιοι επίτροποι έχουν μπροστά τους μια ακρόαση από δύο ή και τρεις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Κάτι που στην ουσία τελικά απομειώνει της, ε, την ικανότητα των αρμοδίων να θέσουν τα κέρια ερωτήματα και να λάβουν ικανοποιητικές απαντήσεις σε σχέση με τις ανησυχίες που θα εκφράσουν. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ε, μια σειρά επίτροποι ε, Πώς θα το πω, υπάρχουν μια σειρά χαρτοφυλάκια όπου τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα διαπλέκονται με έναν συγκεχημένο τρόπο με ζητήματα δημοσιονομικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και αυτό δημιουργεί μια δυσαρέσκεια ακόμη και εδώ στις, ε, στις ε, αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές που καλούνται να ασκήσουν τον κοινοβουλευτικό τους έλεγχο. Και να σας πω ότι εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας εσάς όλους, έχω εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου σε όλες τις επαφές που είχα με τους, με τους οριστέντες επιτρόπους και πρόκειται για τους επιτρόπους που θα έρθουν εδώ για να αντιμετωπίσουν τις ερωτήσεις σας και κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι τους για να απαντήσουν με ικανοποιητικό τρόπο. Έχω κάνει το σχόλιο αυτό και το, το παράπονο αυτό στην ίδια την κυρία Φόντερ Λάιεν, λέγοντάς ότι ο σχεδιασμό αυτός τη Νέα Επιτροπή θα, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο τώρα στην αρχή στις ακροάσεις, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίω όσον αφορά την άσκηση των ε, ελεγκτικών μα αρμοδιοτύπων, προκειμένου να λογοδοτούν οι επίτροποι για τα θέματα που εμπίπτουν στι αρμοδιότητε του. Βεβαίως ε, βλέπω ότι η κυρία σας, σας θέλει να, να, να, πει κάτι ακόμη. Και... Πρόεδρε, μόνο να σας πω και στο Σαλέχος ότι ε, αν γίνουν ε, όλα αυτά θα είναι κρίμα να μην έχουμε την κυρία Γουίδεκομ εδώ στην ε, Επιτροπή μας στο μέλλον. I see your meaning. Α, κατάλαβα που το πάτε λέει ο Πρόεδρος. Να, ναι, σας χάρισε και χαμόγελο. Πάντως, μπράβο, μπράβο για το χιούμορ σας. Σας κύριε, λέω. Τέλος πάντων τώρα να ολοκληρώσουμε. This discussion of us has raised all of the issues. Τα συζητήσαμε όλα, όλα αυτά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, όπως ε, είπα και το είπα σε όλους, μας κάνουν να είμαστε η πιο πολυάσχολη επιτροπή, να έχουμε τις ε, ευρύτερες αρμοδιότητες όλων. Εμείς είμαστε η Επιτροπή Βαριών Βαρών όσον αφορά την ε, νομοθεσία που κάνει το Κοινοβούλιο. Ασχολούμαστε με την προστασία του ιδιωτικού βίου, την προστασία των δεδομένων, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, που είναι οι βασικοί πυλώνες της ε, Ευρώπης. Την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, εσωτερικές υποθέσεις και θέματα ασφαλείας, αστυνομική συνεργασία, την πολιτική, τη στρατηγική ασφαλείας, την αντιμετώπιση του ισορικού εγκλήματος, ε, ασχολούμαστε με την ε, ποινική νομοθεσία, με τα δικαιώματα σχετικά με τη δικονομία, ε, ασχολούμαστε επίσης με το πώς θα υπάρχουν δίκες, δίκες και πάνω από μία φορά έτσι έχουμε προσφύγει και με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με επιτυχία πάνω από μία φορά. Επίσης ασχολούμαστε και με τη δικαστική συνεργασία, ε, κάτι που έχει ω θεμέλιο την αμοιβαία αναγνώριση, αμοιβαία εμπιστοσύνη σε σχέση με τι δικαστικέ αποφάσει. Όλα αυτά, όλα μαζί μα κάνουν την Επιτροπή με τι ευρύτερε αρμοδιότητε. Ευρύτερε σε σχέση με όλες τις άλλες και αυτό αφορά το πόσα χαρτοφυλάκια, πόσους επιτρόπους καλύπτουμε. Ε, γι' αυτό και στην προηγούμενη θητεία είχαμε επαφές με τόσο πολλούς και επίσης έχουμε επαφές με όλες τις κοινοτικές υπηρεσίες σε σχέση με δικαιοσύνη και ασφάλεια. Μιλώ για τουλάχιστον εννέα σχετικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες μας ε, και έχουμε επαφές τακτές. Στην προηγούμενη θητεία είχαμε αντιπρόεδρο που είχε αναλάβει Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή που είχαν λάβει το κράτο δικαίου, τον κύριο Τίμερ μα, είχαμε για τα εσωτερικά τον ε, κύριο Βραμόπουλο, είχαμε την κυρία Γιουρόβα, είχαμε τον Τζούλιαν Κίνγκ και στην επόμενη επιτροπή θα έχουμε τον αντιπρόεδρο που θα ασχολείται με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Θα έχουμε ε, σχετικά με τα δικά μας, την κυρία Γιουρόβα για ευρωπαϊκέ ε, αξίε και διαφάνεια, την, τον κύριο ε, renders για την δικαιοσύνη και για εσωτερικές υποθέσεις την, ε, την κυρία, τον κύριο Γιωχάνσον αλλά επίσης σχετίζονται οι μας και με άλλα χαρτοφυλάκια άλλων υποψηφίων επιτρόπων. πρόσταση του ιδιωτικού βίου που βρίσκεται σε κάποιο ε, χαρτοφυλάκιο και θα χτυπήσουμε και αυτόν τον Επιτρόπο την ε, ε, πόρτα. κατά πολέμηση του ξεπλήματο χρήματο μέσω του ποινικού δικαίου, χρηματοδότηση των τρομοκρατών, αυτά έχουν καλυφθεί από το χαρτοφυλάκιο του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκη που έχει αναλάβει τα οικονομικά. Ενώ στην αρχή ήταν θέματα μόνο ποινικού δικαίου, και αυτά ήταν δική μας αρμοδιότητα. Άρα θα πρέπει να έχουμε κοινέ αρμοδιότητες. Άρα έχουμε λίγο το περιθώριο λιγμών, κοινέ αρμοδιότητες με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και αυτό αφορά και τις ε, ακροάσεις. Ελπίζω όσοι στήσαμε σήμερα θα βοηθήσουν τους συντονιστές. Οι από συντονιστές εκείνοι θα αποφασίζουν για την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων ή τέλο πάντων των θεμάτων που θα τεθούν από κάθε, προς κάθε ε, πολιτικό κόμμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης για τις ερωτήσεις προς τους ε, ε, επιτρόπους θα έχουμε 25 ερωτήσεις. Ε, αυτό είναι εξάρτητο πόσες θα είναι οι συνάνομαδες επιτροπές. Έτσι θα εξετάσουμε τους υποψηφίους επιτρόπους, η τις υποψηφίους, επομένως έχουμε 25 ερωτήσεις ε, θα κατανεμηθούν σε όλες τις πολιτικές ομάδες ε, ανάλογα με το μέγεθος κάθε πολιτικής ομάδας ε, μέχρι πέντε στις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες και μικρότερες ε, μία ερώτηση. Άρα οι συντονιστές θα έχουν το σπουδαίο έργο να διατυπώσουν την ερώτηση και επίσης να οριστεί ποιοι βουλευτές θα λάβουν τον λόγο να εκφωνήσουν την ερώτηση. Και ξαναλέω, ελπίζω ότι όσα είπαμε θα βοηθήσουν τους συντονιστές. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Να, για μια φορά κάναμε ελεύθερη, χαλαρή συζήτηση και καλύψαμε όλα αυτά τα θέματα που θέλαμε. Τώρα, για να κλείσω, να σας πω τον ρόλο της Επιτροπής μας, γιατί πάρα πολύ σημαντικό. Την πολιτική κατά των δεσμενών διακρίσεων. Σε όλα τα θεσμικά όργανα και από όλα τα θεσμικά όργανα. Μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα η ισότητα. Να τα απολαύουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Είμαστε κατά, κατά των δυσμένων διακρίσεων, κατά του στιγματισμού, κατά των προκαταλήψεων. Ε, εθνική προέλευση, ε, θρησκεία, γλώσσα οποιασδήποτε ιδιότητα δεν θα πρέπει να είναι στόχος της μενινούς διάκρισης. Όλα θα μας ενδιαφέρουν και καλά κάνουμε. Αυτό θέλουμε. Ίσα δικαιώματα για όλους. Και γι' αυτό και έχουμε και το σχετικό καινούριο χαρτοφυλάκιο. Η Ελένα Ντάλι το έχει αναλάβει. Η Ελένα Ντάλι από την Μάλτα. Άρα έχουμε να χειριστούμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα τελευταία μου σκέψη ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την αρχή της διαδρομής ότι αυτά μέσα στα θέματα όχι μόνο είναι πάρα πολύ απαιτητικά και έχουμε κάποιες περίπλοκες διαδικασίες να ε, περάσουμε για να καταλήξουμε σε κάποιο νομοθέτημα, την πρώτη ανάγνωση, τη δεύτερη ανάγνωση, τις ε, συνδιαλλαγές, κάποιους ε, τριμερείς διαλόγους που κρατάνε καμιά φορά χρόνια. Τα έχουμε δει και τα ξαναδεί όλα αυτά και θα τα ξαναδούμε. Είναι βέβαια. Όχι μόνο τα θέματα είναι δύσκολα, αλλά είναι και διχαστικά από πολιτικής πλευράς. Άρα να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε. Έχουμε και πολλές αρμοδιότητες, αλλά και καυτές αρμοδιότητες. Κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας, ούτω ώστε να έχουμε αλληλοσεβασμό, εγγύηση ελευθερίας λόγου, αλλά επίσης σίγουρα θα υπάρξουν και προστριβές. Επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα. Κάθε πολιτική ομάδα δικαιούται να τοποθετηθεί και επίσης θα πρέπει να ακούσει και τα αντεπιχείρηματα. Οπότε, σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Και προχωράμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μου είπαν ότι έχουν έρθει συνέχεια τηλεόραση για να έρθουν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Πες τη ξέρω πώς λέγεται το κανάλι αυτό, pisterakol.hu. Άρα είναι ουγγρικό κανάλι. Ναι, ναι. Ουγγρικό. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα του ε, επιτρέψουν να μπουν στην αίθουσα για να τραβήξουν αυτά τα πλάνα. Υπάρχει ένσταση. Όχι, καλώ. Πάμε ακόμα στο επόμενο σημείο τη μερική διάταξη που είναι ο κανονισμό VIS. Σα υπενθυμίζω. Έχουμε ψηφοφορίες που ξεκινούν στις 6. 6. Άρα, να αντέξετε μέχρι τότε και σύνεργα. Και θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μπαρτόλου, και θα επιστρέψω το συντομότερο. Allora, Συνάδελφοι, όσο αφορά τώρα αυτό το σύστημα VIS, ήδη οι προσπάθειε και εργασίε έχουν αρχίσει πριν τι ευρωεκλογέ και θα συνεχιστεί η συζήτηση ε, να εμβαθύνουμε στο θέμα, οπότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ραντζέλ. Uh, Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο τίτλος αυτού του σημείου της σημερινής διάταξης μάλλον μας μπερδεύει. Γιατί, όπως είπατε, το Κοινοβούλιο έχει κάνει την ανταλλαγή απόψεων εσωτερικά στην προηγούμενη θητεία, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και έχει αποφασίσει τη θέση του. Η Ολομέλεια εγκρίνει τη θέση μας για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν επαναλαμβάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ για ανταλλαγή απόψεων με τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό ναι. Αλλά δεν διαπραγματευόμαστε ακόμη. Χρειαζόμαστε ακόμη την έγκριση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Στη ψηφοφορία που θα γίνει σήμερα σε λίγες ώρες. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας. Γι' αυτό και εγώ θα επαναλάβω σε γενικές γραμμές, τις βασικές γραμμές της θέσης του Κοινοβουλίου, για τις οποίες θέλουμε την εντολή να διαπραγματευτούμε. Καταρχήν θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στα σύνορά μας και γι' αυτό μιλάμε για τις θεωρήσεις διαβατηρίου μακράς διαρκείας και ιδιαίτερα τις χρυσές βίζες, τις οποίες συμπεριλαμβάνουμε στο σύστημα και αυτή η αλλαγή θα προστατεύει καλύτερα τα σύνορά μας και θα διασφαλίζει και τα δικαίωμα των ε, όσων ε, διαμένουν μακροπρόθεσμα και θα διευκολύνει την ε, μετακίνηση. Δεύτερον, Θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και γι' αυτό ε, δίνουμε τη δυνατότητα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, να γίνεται και ε, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως ότι θα ισχύσουν απόλυτα αυστηρές προδιαγραφές και διασφαλίσεις υπέρ της προστασίας των παιδιών. Τρίτον, θέλουμε να έχουμε μια λειτουργική αρχιτεκτονική και τεχνικά και νομικά. Επομένως, η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι πρέπει να ανακαλέσουμε την πρόταση του Συμβουλίου για το VIS και να ε, ευθυγραμμιστεί το σύστημα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα όμως θα αυξάνεται, η ζήτηση θα αυξάνεται και γι' αυτό θέλουμε τα υψηλότερα δυνατόν πρότυπα όταν μιλάμε για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτού του μέτρου. Τέταρτο σημείο, πλην όμως όχι έσχατο, θέλουμε να υλοποιηθεί εγκαίρως και με βάση τον προϋπολογισμό. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων και προθεσμίες για την υλοποίηση των νομοθετικών μέτρων. Από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι πολύ συχνά, δυστυχώς, ξεφεύγουμε από τον προϋπολογισμό και από τις προθεσμίες λόγω διαφόρων προβλημάτων με τα συστήματα πληροφορικής. Βάζουμε λοιπόν μια προθεσμία δύο ετών κατά μέγιστο για την μεταρρύθμιση αυτή, για να αρχίσει να λειτουργεί πλέον αυτή η μεταρρύθμιση. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή είναι η εντολή που θα έχουμε για τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο, εφόσον έχουμε θετική ψήφο σας σήμερα το απόγευμα. Με τους σκιώδεις εισηγητές θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις ε, όλων και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που συνόψισε τη δουλειά που κάναμε κατά την προηγούμενη θητεία. Και την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση και ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για όλες τις πολιτικές ομάδες που μπόρεσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι όντως ψηφίστηκε το θέμα αυτό στην προηγούμενη θητεία και έπρεπε να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό το οποίο είχε ψηφιστεί, αλλά είχαμε καθήκον να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις. Επίσης, οι στόχοι όπως τους ανέφερε ο εισηγητής με βρίσκουν σύμφωνο. και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την υλοποίηση με σαφές χρονικό πλαίσιο και προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να εκφράσω την ανησυχία μου για κάτι. Δεν ε, θέλω να ε, εκφράσω αμφιβολίες για την εντολή που μας είχε δοθεί, αλλά την προηγούμενη φορά που εξέφρασε το Κοινοβούλιο τη θέση του ήταν πολύ κοντινές οι απόψεις και αυτό αφορά την προστασία των παιδιών. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα γιατί θυμάμαι και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει πριν από χρόνια για το θέμα αυτό όταν εφαρμόστηκε το VIS. Οι τεχνικοί πυρογνώμονες φαίνεται ότι άλλαξαν γνώμη τώρα, γιατί πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαν ότι τα αποτυπώματα, δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών κάτω από 12 ετών δεν μπορούσε να γίνει, ούτε τεχνικά. Δεν μας έδινε βαθμό αναγνώρισης ικανοποιητικό και δεν θα βοηθούσε φαίνεται ότι μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξαν οι τεχνικές δυνατότητες και αυτό μου δημιουργεί έκπληξη. Επίσης δεν είμαι πεπισμένος για τα οικονομικά επιχειρήματα. Είδα κάποια στοιχεία, εκατομμύρια θεωρήσεις δίδονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών και άρα ε, αυτό συνδέεται με την ε, παράνομη διακίνηση παιδιών. Με ανησυχεί πάρα πολύ η παράνομη διακίνηση παιδιών και εμένα όπως και όλους μας στην αίθουσα αυτή, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι τα παιδιά αυτά που είναι θύματα διακίνησης ήταν παιδιά τα οποία ήρθαν νομίμως με θεωρήση διαβατηρίου από μια νόμιμη διέλευση συνόρων. Πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά διακινούνται παράνομα μέσω των παράνομων οδών μετανάστευσης στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα σημεία που θέλω να θέσω προς συζήτηση. Και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και να βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα έχει το λόγο. Η κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή επίσης. Τον ευχαριστώ για όσα έκανε στο Στρασβούργο και απλώ τον Πρασίνων θέλω να πω ότι εμεί υποστηρίζουμε την θέση που δημοσιεύθηκε στην προηγούμενη θητεία. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ αρνητικό το ότι δεν αποσπάσαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, όμως θεωρούμε ότι είναι θετική η συζήτηση που έγινε, οι επαφές που έγιναν και όσα είπαμε στην τελευταία ε, συνάντηση που συζητήσαμε το όριο ηλικία για λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ελπίζουμε ότι αυτό θα ληφθεί αυτή στο μέτρο ε, και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα τα πάμε καλύτερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος, και τώρα Δώσουμε το λόγο σε όποιο συνάδελφο θέλει το λόγο. Σε μια ελεύθερη ζήτηση. Ράντα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά Η κατάσταση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά κενά νομικής φύσεως. Οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν επαρκείς μηχανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα συστήματα με πολύ ξεχωριστούς όμως και ε, επιμέρους στόχους και ε, το κάθε σύστημα διατηρεί στα πλαίσια του τις διάφορες πληροφορίες χωρίς δυνατότητα σύγκρισης των πληροφοριών του ενός συστήματος με τις πληροφορίες ενός άλλου ε, με τις πληροφορίες ενός άλλου συστήματος. Γι' αυτό και χρειάζεται να προχωρήσουμε στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας ακριβώς για να μπορέσουμε να συνδέσουμε πληροφορίες από το σύστημα ε, πληροφοριών θεωρήσεων, για παράδειγμα, με τις πληροφορίες από το σύστημα Schengen, και τα άλλα συστήματα, ώστε όταν ένας συνοριοφύλακας ελέγχει κάποιο διαβατήριο να μπορεί να αναζητεί πληροφορίες σε όλα αυτά τα συστήματα. Έχει ήδη γίνει μια τέτοια πρόταση και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ξεκινήσει και η σχετική ε, διαθεσμική διαπραγμάτευση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τη δυνατότητα στους αξιωματούχους των αρχών επιβουλής του νόμου να χρησιμοποιήσουν ε, όλες τις πληροφορίε που έχουμε στη διάθεσή μας ε, στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιομετρικά και άλλα, για να μπορεί να επαληθεύει την ταυτότητα του κάθε εισερχόμενου ατόμου. Για να γίνουν όμω όλα αυτά, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν υψηλή ποιότητας πληροφορίε. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία και η παράνομη μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει η κυρία Νικολσονόβα. Ευχαριστώ πολύ. Ως σκιώδης εισηγήτρια να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση αυτή γιατί θεωρώ ότι θα βελτιώσει σημαντικά το σύστημα VIS. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μετανάστευση ήταν σημαντικότατα ζήτημα που απασχόλησε την προηγούμενη θετία και δεν βρήκαμε τις ιδανικότερες δυνατές λύσεις. Όμως συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια ιδίως στα εξωτερικά σύνορα και από αυτή την άποψη πραγματικά χαιρετίζω την πρόταση. Έχω όμως ε, και κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Ακούστηκαν ήδη κάποιες από αυτές. Πρώτον, σε αντίθεση με το Συμβούλιο, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την εφαρμογή των τροποποιήσεων των αλλαγών στον φάκελο αυτό. Δεν συμφωνώ να μείνουν ανοιχτά τα πράγματα όπως προτείνει το Συμβούλιο. Δεύτερον, μόλις ξεκινήσει το σύστημα να λειτουργεί και για άδειε παραμονής και μακροχρόνιας διαμονή θα πρέπει να ορίσουμε και συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης δεδομένων. Όπως οι χώρες μας έχουν αρχεία και μητρό για εμάς, τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί να μην έχουν πληροφορίε και για υπηκόου τρίτων χωρών, όταν τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στην επικράτεια των χωρών μας. Τέλος, δακτυλικά αποτυπώματα παιδιών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια συζήτηση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η μελέτη του Κοινού Κέντρου Έρευνας αποδεικνύει ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από άτομα ηλικίας 6 έως 12 ετών είναι εφικτή και μάλιστα είναι καλύτερης ποιότητας από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων άνω των 65 ετών. Χρειάζεται βεβαίως να εκπαιδευτούν εκείνοι που χρειάζεται να λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την μεταβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών. Τέλος, η έκθεση της Κομισιόν για την καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων αναφέρει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις έως 2.000 παιδιά το χρόνο γίνονται θύματα διακίνησης στον χώρο Σέγγεν και μάλιστα 25% αυτών των παιδιών έχουν περάσει μέσα από το σύστημα των θεωρήσεων. Άρα έχουμε τους αριθμούς τους, έχουμε τα ονόματά τους και τα βιομετρικά τους δεδομένα. Πληροφορίες που τις έχουμε, άρα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως είναι ο κανονισμός για την ε, δημιουργία των ε, καρτών άδειας παραμονής, αναφέρει ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι υποχρεωτική για άτομα και παιδιά άνω των 6 ε, ετών. Όλα αυτά προβλέπονται αλλά δεν εφαρμόζονται πάντοτε. Η Δανία, για παράδειγμα, προβλέπει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμένων από παιδιά 6 ετών και άνω. Άλλε χώρες, όπως η δική μου χώρα, για παράδειγμα, η Σλοβακία, ξεκινούν από την ηλικία των 10 στην εκτίμηση, της, στην εκτίμηση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα αναφέρει ότι από τη σκοπιά ε, των δικαιωμάτων των παιδιών η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων μαζί με τη βελτιστοποίηση άλλων πληροφοριακών συστημάτων όπως είναι το SIS-2 μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό χαμένων παιδιών και να διευκολύνουν τη διαδικασία επανένωσης οικογενειών. Και αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο και για τα παιδιά στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταναστευτικής και προσφυγικής κατάστασης. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, να πω ότι για να καταπολεμηθούν όλα τα είδη σοβαρού εγκλήματο, η διαθεσιμότητα δακτυλικών αποτυπωμάτων και παιδιών κάτω των 12 ετών έχει προστιθέμενη αξία, ακριβώς γιατί μπορούν να ελέγχονται αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα ε, σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που έτσι κι αλλιώ και ήδη τηρούνται. Και το λέω αυτό ότι θα πρέπει να γίνεται αυτή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά κύριο λόγο για να προστατεύονται τα ίδια τα παιδιά. Κύριος Μπρισμόν. Στα παλάντο. Α, ο Λέει; I'm uh, Πρόεδρε, δεν δε ζήτησα το, το λόγο. Συγγνώμη, κάποιο λάθος έχει γίνει, λέει η κυρία Μπρικμόντ. Το και vuole intervenire. Στέλνει κάποιο άλλο το λόγο. Όχι, κανείς. Οπότε. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Γκρός. Uh, Ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ρανσέλ, που συνέχισε να είναι επικεφαλής ε, αυτής της διαδικασίας, αυτού του φακέλου και στις διαπραγματεύσεις. Ξέρετε ότι μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό το θέμα αυτό. Θέλω σε αυτή τη φάση να ανακοινώσω ότι με το νέο σύστημα θεωρήσεων θέλουμε να άρουμε συγκεκριμένα προβλήματα και ελλείψεις που υπήρχαν και να δώσουμε στις αρχές μας τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτελέσουν και να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους με το σωστό τρόπο. Το σύστημα θεωρήσεων μαζί με το αίτιας και το σύστημα εισόδου-εξόδου αποτελούν τμήματα μια ενιαία πλατφόρμα που αφορά του υπηκόου τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό τα συστήματα αυτά να είναι συγχρονισμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν χαιρετίζει την υποστήριξη που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το βασικό στόχο τη πρότασή μα και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με του συνομοθέτε στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πολλά από τα ζητήματα που ο εισηγητή και οι άλλοι ευρωβουλευτέ έθεσαν σήμερα. Ελπίζουμε βεβαίως να είμαστε σε θέση γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση αυτή και να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της ασφάλεια και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ασφαλέστερη ένωση προ όφελο των πολιτών μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Φινλανδικής Προεδρίας, θέλω να πω ότι η Προεδρία έχει δεσμευθεί ότι το θέμα αυτό θα το προωθήσουμε κατά την Φινλανδική Προεδρία. Συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία που ανέφερε ο εισηγητής ο κύριος, ο κύριος ίσως ε, να τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά σε κάποια σημεία, αλλά τις βασικές προτεραιότητες τις συμμεριζόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν καλά για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα με στόχο την ασφάλεια των συνόρων, την ασφάλεια των παιδιών μας. και εκ μέρους της Φιλανδικής Προεδρίας θέλω να πω ότι κατανοούμε ότι το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου θα πρέπει να είναι μια συμβιβαστική λύση που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σημεία τα οποία αναφερθήκαν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ. Και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Τσουχοντάρου. Η έκθεση αυτή πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Υπάρχουν κάποιες ε, λεπτομέρειες που ελπίζω ότι θα διευκρινιστούν κατά τις διαπραγματεύσεις και θέλω να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι συμμετείχαν. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι έχει γίνει πολλή δουλειά με ανοιχτό πνεύμα και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε βελτίωση της ασφαλείας μας και σε λιγότερα τραγικά συμβάντα. Ευχαριστώ. Μήπως θέλει να ολοκληρώσει κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για όσα είπαν και σας επαναλαμβάνω ότι είναι καλά τα νέα το ότι προτίθεται Συμβούλιο και Κομισιόν να διαπραγματευθούν Δεν χρειάζεται προς το παρόν κάποιο σχόλιο. Ελπίζω η ψηφορία θα είναι θετική και θα αρχίσουμε τη δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο, το οποίο αφορά το έγγραφο εργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής με θέμα. Ανάλυση μέτρων δίμευσης που δεν βασίζονται σε καταδίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ το έγγραφο το οποίο προετοιμάσαμε για τη δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Η δίμευση και η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντικά στοιχεία για την καταβολέμηση ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Το έγγραφο το οποίο θα σας παρουσιάσω για τη δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη βασίζεται στη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του, του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μετά την οδηγία για τη δίμευση του 2014. Ίσως να θυμάστε ότι οι συνομοθέτες είχαν ζητήσει τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύει τα μέτρα δίμευσης ε, κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έγγραφο είναι το πρώτο βήμα στην ανάλυση της Επιτροπής. Η επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα αυτό θα προκύψει μέσω μιας έκθεσης την οποία ε, ε, θα στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας για τη Δήμευση. Αυτή θα είναι η επίσημη απάντηση στην κοινή διακήρυξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η ακριβή ημερομηνία για την παρουσίαση αυτής ε, της έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασιστεί από τη νέα Επιτροπή, από το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων. Πάντως θα είναι μέσα στο πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο του 2020. Έχω προετοιμάσει μία σύντομη παρουσίαση για να σας αναφέρω ποιο είναι το υπόβαθρο, τι νομοθετικές διατάξεις έχουμε ήδη και να περιγράψω και τα ευρήματα της δικής μας έκθεσης για τη δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Καταρχήν, για το γενικό πλαίσιο, το οργανωμένο έγκλημα είναι μια δραστηριότητα που κινείται κυρίως ε, με σκοπό τα κέρδη. Το κέρδος είναι αυτό που κάνει τις εγκληματικές οργανώσεις να κάνουν αυτό που θέλουν. Από το Ινστιτούτο Transcrime υπολογίζεται ότι τα έσοδα είναι 110 δισεκατομμύρια ευρώ από το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ε, νομίζω χαμηλές οι εκτιμήσεις αυτές. Ε, τα προϊόντα εγκληματικών ενεργειών είναι 3,6% του συνολικού ΑΕΠ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα προϊόντα του εγκλήματος και αυτά τα κέρδη επενδύονται από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις είτε για να διαδώσουν περαιτέρω τις ε, δραστηριότητές τους είτε για να αρχίσουν να μπαίνουν στην νόμιμη οικονομία. Η οργανωμένη εγκληματικότητα λοιπόν αποτελεί απειλή και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός ο μηχανισμός ε, για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, το να μπορέσουμε να πάρουμε από τις εγκληματικές οργανώσεις ε, τα χρήματα αυτά που είναι προϊόντα του εγκλήματος. Είναι όμως πολύ πολύπλοκη αυτή η διαδικασία στην πράξη. Διότι οι εγκληματικές οργανώσεις προσπαθούν να αποκρύπτουν τις ε, χρηματοοικονομικές ροές και είναι δύσκολο για τις αρχές επιβολής του νόμου ε, να βρουν τις σχέσεις μεταξύ ε, εγκληματικών δραστηριοτήτων και κερδών τα οποία έχουν προκύψει από αυτές τις δραστηριότητες. Τα νομικά καθεστώτα, λοιπόν, τα νομικά συστήματα που επιτρέπουν την ε, δίμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς καταδίκη είναι μέσα τα οποία έχουν ε, αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που, υπάρχουν σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες και τα κέρδη αυτών. Η δίμευση παραδοσιακά βασιζόταν σε μοντέλα που βασίζονται σε αποφάσεις καταδικαστικές. Οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία που θα του δώσουν τη δυνατότητα να δημεύουν προϊόντα εγκλήματος ε, σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Μόνο 1% των κερδών του οργανωμένου εγκλήματος δημεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανάλυση μας λοιπόν προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα διάφορα μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διάφορα κράτη-μέλη και στην ανάλυση αυτή εμπνευστήκαμε από ένα οδηγό του δικτύου Camden, το, είναι το δίκτυο Karin, που ανέπτυξε αυτόν τον οδηγό το 2015 με μια τυπολογία με τέσσερα μοντέλα. Και αυτή η ταξινόμηση μας βοηθά να κατηγοριοποιήσουμε τις προσεγγίσεις των κρατών μελών. Εμπνευστήκαμε από τα μοντέλα αυτά και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι υβριδικά αυτά τα μοντέλα. Δηλαδή το κάθε μοντέλο συμπεριλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία και από άλλα μοντέλα, δεν είναι αμυγή μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο είναι η δίμευση που θα την αποκαλούσαμε παραδοσιακή δίμευση που βασίζεται ε, σε μέτρα που δεν συμπεριλαμβάνουν καταδικαστική απόφαση. Όταν η δίμευση δεν είναι εφικτό να γίνει με βάση μια τελική καταδικαστική απόφαση, παραδείγματο χάρη για λόγους όπως το ότι έχει αποβιώσει ο ύποπτος ή ότι έχει διαφύγει ο δράστης, έχει φύγει από τη χώρα και δεν μπορούμε να τον βρούμε. ή γιατί το δικαστήριο θεωρεί ότι ε, δεν μπορεί να διωχθεί ο δράστης λόγω ασυλίας ή λόγω της ε, ψυχικής του υγείας ε, ή ηλικίας ή οτιδήποτε. Το δεύτερο μοντέλο τώρα είναι η διευρυμένη, η εκτεταμένη δίμευση που επιτρέπει τη δίμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με το έγκλημα για το οποίο διώκεται ο δράστης. Επομένως, η εντολή δίμευσης μπορεί να επεκταθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία ε, του δράστη το τρίτο μοντέλο είναι η διαδικασία η εμπράγματη, η διαδικασία in rem, που δεν είναι διαδικασία κατά του ατόμου, αλλά κατά των εμπράγματων στοιχείων. Και το τελευταίο μοντέλο, το τέταρτο μοντέλο, ε, είναι το μοντέλο αδικαιολόγητου πλουτισμού, δηλαδή συγκρίνει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει ένα άτομο έναντι του εισοδήματος το οποίο έχει δηλώσει, προσπαθώντας να προσδιορίσει τη διαφορά μεταξύ των δύο και προσπαθεί να βρει μία ε, σχέση έστω και έμεση με το κύριο αδίκημα. το νομικό πλαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την ανείχνευση, για την δέσμευση και δίμευση περιουσιακών στοιχείων είναι μία απόφαση του Συμβουλίου για ε, ένα δίκτυο γραφείων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στα κράτη-μέλη και βοηθούν την αστυνομία να εντοπίσει περιουσιακά στοιχεία. Επίσης υπάρχει η οδηγία για τη δίμευση που εγκρίθηκε το 2014 που προσπαθεί να εναρμονίσει τα μέτρα δέσμευσης και δίμευσης σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλουμε έκθεση για το πώς εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία. Ένας νέος κανονισμός εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2018 για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, εντολών για δέσμευση και δίμευση από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίοδος για την ε, μεταφορά σε εθνικό δίκαιο είναι μέχρι του χρόνου το Δεκέμβριο του 2020. Επίσης πρόσφατα εγκρίθηκε μια οδηγία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες που βοηθά τις αρχές επιβολή του νόμου, θα τις βοηθά όταν μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο, να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία, δίνοντάς τους άμεση πρόσβαση στα συστήματα κεντρικών λογαριασμών, στα συστήματα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Τον Αύγουστο του 2021 λύγει η περίοδος για την μεταφορά αυτής της οδηγίας σε εθνικό δίκαιο. Η οδηγία για τη, για τη δίμευση που εγκρίθηκε το 2014 περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα δίμευσης μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Στο κλασικό μοντέλο, στο κλασικό μοντέλο δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη για τι περιπτώσει που ανέφερε που μπορεί να έχει αποβιώσει ο δράστη ή για λόγου ασθενεία κλπ. Υπάρχει μια διάταξη όπως και στην, στην εκτεταμένη δίμευση και υπάρχουν ε, και διατάξεις ε, για δίμευση ισχύρας τρίτου με κάποιες διασφαλίσεις για την δέσμευση και για την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το άρθρο 4 είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε τώρα με τα μικρά γράμματα στην οθόνη, μπορείτε όταν θα πάρετε την παρουσίαση να το δείτε. Είναι μια διάταξη που μιλά για μέτρα δίμευσης μη βασιζόμενη σε σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο όταν η ποινική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί ο κατηγορούμενος είναι ασθενής ή έχει διαφύγει. Αυτοί οι δύο λόγοι δίνονται. Τα κράτη-μέλη πρέπει στις, ε, στην εθνική τους νομοθεσία να έχουν μέτρα για δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Στο άρθρο 5 η οδηγία παρουσιάζει το μοντέλο εκτεταμένης δίμευσης, όπως σας το παρουσίασα προηγουμένως, επιτρέπει στα κράτη-μέλη, στο εθνικό τους δίκαιο, να έχουν μια δυνατότητα η δίμευση να καλύπτει ε, περιουσιακά στοιχεία που δεν συνδέονται με το έγκλημα για το οποίο διώκεται ο δράστης εάν θεωρείτε ότι, το, ότι τα περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από την εγκληματική δραστηριότητα. Στο άρθρο 6 έχουμε ε, δίμευση που σχετίζεται με τρίτους. Επιτρέπεται η δίμευση λοιπόν περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον όταν έχει μεταφερθεί το περιουσιακό στοιχείο σε τρίτους για την αποφυγή της δίμευσης. Εδώ βλέπετε την κοινή διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν ε, εγκρίθηκε η οδηγία για τη δίμευση. Οι Ευρωπαίοι Συνομοθέτες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το συντομότερο δυνατόν και να λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των νομικών παραδόσεων και των συστημάτων των κρατών μελών, να αναλύσει την βιωσιμότητα και τα πιθανά ωφέλη από την εισαγωγή νέων κοινών κανόνων για τη δίμευση. Αυτό κάναμε τώρα λοιπόν. Σαν ένα πρώτο βήμα εξετάσαμε την κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη αναλύουμε και παρουσιάζουμε τα συστήματα των κρατών μελών και τα όσα έχουν κάνει τα κράτη-μέλη έκτοτε. Αυτό το οποίο είδαμε από την ανάλυση αυτή που κάναμε είναι ότι πολλά κράτη-μέλη, 25 κράτη-μέλη συγκεκριμένα, όλα τα κράτη-μέλη εκτός της Βουλγαρίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή, βασίζονται κατά κύριο λόγο στο κλασικό μοντέλο της δίμευσης μη βασιζόμενης σε καταδίκη. Δηλαδή σε περίπτωση αποβιώσαντος ε, δράστου ή διαφυγόντος δράστου. 26 κράτη-μέλη έχουν την, ε, το σύστημα εκτεταμένης δίμευσης, όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή εκτός της Ελλάδας και της Ιρλανδίας. Επίσης, 13 κράτη-μέλη έχουν κάποια μορφή διαδικασιών ε, για δικαιολόγητο πλουτισμό που συγκρίνουν τα περιουσιακά στοιχεία ενός ατόμου και την φορολογική του δήλωση. Αυτό το έχουν επιπροσθέτως. Τρία κράτη-μέλη βασίζονται μόνο σε αυτό αυτές τις διαδικασίες αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Υπάρχουν όμως πολλά υβριδικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το κλασικό μοντέλο δίμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη, υπάρχουν πολλές διαφορές στα κράτη-μέλη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτών των μοντέλων. Οκτώ κράτη-μέλη καλύπτουν τις περιπτώσεις ασθένειας ή διαφυγής. Τέσσερα κράτη-μέλη καλύπτουν και το θάνατο και άλλα τέσσερα κράτη-μέλη αποκλείουν την αιτία θανάτου. Επτά κράτη-μέλη καλύπτουν μόνο την ασθένεια ή διαφυγή. Επτά κράτη-μέλη καλύπτουν θάνατο, ασθένεια ή διαφυγή. Δύο κράτη-μέλη, η Δανία και η Ελλάδα, καλύπτουν μόνο την περίπτωση θανάτου. Ένα κράτος μέλος, η Γερμανία, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τις οποίες δεν είναι εφικτή η δίμευση στις ποινικέ ε, υποθέσεις και έχει ένα πρόσφατο σύστημα η Γερμανία για ε, έχει υιοθετήσει ένα πρόσφατο σύστημα για τη δίμευση. Και ένα κρατοσμέλος, η Ρουμανία, καλύπτει μόνο την περίπτωση ασθένειας του κατηγορουμένου ή υπόπτου. Όπως βλέπετε υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να συμπεράνουμε με βάση την ανάλυση που κάναμε βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης μετά την έγκριση της οδηγίας για τη δίμευση. Πλην όμως υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει και πέραν των ελάχιστων απαιτήσεων για τα μέτρα δίμευσης μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Έχουν αναπτύξει περισσότερο τα μοντέλα αυτά. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι τα συστήματα δίμευσης μη βασιζόμενα σε καταδίκη μπορούν να αποδώσουν πολλά. Δεν έχουμε όμως ακόμη αρκετά δεδομένα για να μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε. Κάποια συστήματα που έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη πληρούν τις απαιτήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τουλάχιστον μέχρι τώρα ε, κανένα από τα συστήματα αυτά δεν έχει καταπέσει σε δικαστήριο. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω και προσβλέπω στην ε, ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στίγελ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, μας κάνει πλάστη σε υπηρεσία σας για αυτά τα μέτρα τέτοιας ε, διαδικασίας δίμευσης χωρίς δηλαδή προηγούμενη καταδίκη. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να λάβει τον λόγο. Ο κ. Ράντεφ, αντιπρόεδρος, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτού του εγγράφου. Πολλέ φορέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει θέσπιση κανόνων, ώστε να υπάρχει ένα στεγανό νομοθετικό πλαίσιο για την ε, δίμευση προϊόντων εγκλήματος. Η δίμευση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 99% των προϊόντων εγκλήματος δεν δημεύονται. Πάντως, η αμοιβαία αναγνώριση των νομοθετημάτων και των σχετικών ενταλμάτων είναι κάτι που έχει αποδώσει στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Οπότε τα κρατημέλη και εν προκειμένου θα μπορέσουν να επεκτείνουν τα όσα ισχύουν ε, και στην ε, δίμευση ισχύρας τρίτου. Βέβαια ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, κάθε εθνικό δίκαιο είναι διαφορετικό από τα άλλα, αλλά είδαμε ότι πάρα πολλά κρατή-μέλη κάνουν μεταρρυθμίσεις και θεσπίζουν μέτρα τέτοια της τέταρτης κατηγορίας όσον αφορά τη, τη δίμευση. Βέβαια ποτέ δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι πρέπει να ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Βουλγαρία. Χρησιμοποιούμε αυτή την τέταρτη κατηγορία μέτρων δίμευσης και έχουμε αποσπάσει αξιολόγο αποτελέσματα τώρα πρόσφατα, αλλά τι θα γίνει στο μέλλον, αυτό θα ρωτήσω Ευρωπαϊκή τώρα πώς θα έχουμε περαιτέρω εναρμόνιση. Επίσης, τι θα γίνει με την τέταρτη κατηγορία μέτρων δίμευσης σε σχέση με την μεταρρύθμιση που έπεται. Κυρία Σίπελ, ναι. Και αυτό το θέμα είναι δύσκολο γιατί νομίζω ότι πολλοί συμπολίτε μας δεν καταλαβαίνουν γιατί πολλές φορές καταδικάζονται κάποιοι εγκληματίες και ταυτόχρονα όμως δεν χάνουν ότι αποκόμψαν από το έγκλημα. Επίσης είναι δύσκολη η υπόθεση αυτή των δημιουργήσεων χωρίς καταδίκη γιατί θα πρέπει να δούμε Πώς δεν θα υπερβάλλουμε στη ρύθμιση. Οπότε συμφωνώ που είπε η Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε ένα στεγανό σύστημα με σεβασμό δικαιωμάτων. Οπότε όλα αυτά θα είναι βέβαια πρόοδο. Τώρα άλλο θέμα. Η δίμευση είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα όμως είναι τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία που δημεύονται. Οπότε μου λένε, το κάθε κράτος μέλος έχει άλλη πολιτική σχετικώς. Δεν ξέρω, ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ισχύει. Όλα αυτά πάνε στο κρατικό προϋπολογισμό. Τι γίνεται, αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα για διάφορους σκοπούς. Έχουμε στοιχεία για το πώς πρέπει με τον τρόπο να το ρυθμίσουμε. Η κυρία Τουγκάρου. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τα όσα μας εξήγησε. Περιμένω να προκύψουν και άλλα για τη συνέχεια αυτή τη διαδρομής, να έχουν περισσότερε πληροφορίες. Δεν έχουμε αρκετέ από κρατών άλλων, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Να γίνει μια πιο σφαιρική ανάλυση και ετησίω 110 δι ευρώ έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοιες πράξεις και μόλις 1% ανακτάται. Κάναμε βήμα πρόοδο, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι υπήρξαν ε, αντίθετες αποκλίνωσες απόψεις για το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Το αρχικό άρθρο 5 της οδηγίας αυτής τελικά αντικαταστάθηκε όλο μαζί από μια πολύ απονευρωμένη διάταξη. Που περιορίζει πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογή τη ρύθμιση, τη δίμευση αυτή. Ρωτώ την Επιτροπή. Θα τολμήσουμε, θα είμαστε πιο εύστοχοι στη ρύθμισή μας, γιατί περισσότερα κράτη-μέλη έχουν το κλασικό μοντέλο. Αχ, στη Ρουμανία, τη χώρα μου, μόνο εν μέρη εφαρμόζεται το πρώτο μοντέλο. Στην Βουλγαρία, που έχει πετυχημένη εφαρμογή του μέτρου και χρησιμοποιεί την αντιστροφή του βάρους αποδείξεως, Αρκεί το να μην υπάρχουν στοιχεία που προέρχεται την περιοχή. Να δούμε τι κάνει η Ιταλία, τι κάνει η Γερμανία, που επιτυχώ συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα. Το 2, 3, 4, α πούμε, που τα ακούσαμε, μα τα παρουσιάσανε. Οπότε, μετά από την ε, σχετική έκθεση τον Οκτώβριο ή αρχές του 2020 μπορούμε κάτι να κάνουμε ούτως ώστε να ενισχύσουμε το πλαίσιο για ε, κλασική δίμευση, αλλά επίσης και να μπορέσουμε να θεσπίσουμε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ωραία. Θα κάνω κι εγώ μια καταληκτική παρατήρηση για το θέμα, αλλά ας ακούσουμε πρώτα τους ε, ευρωβουλευτές. Η κυρία Στρίκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ως πράσινοι υποστηρίζουμε πλήρως βεβαίω ε, την ιδέα ότι οι εγκληματίε δεν θα πρέπει να ωφελούνται από τα εγκλήματα που διαπράττουν. Και θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή για την εποπτεία που μας παρέχει σχετικά με τι διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούνται σε εθνικό επίπεδο, ε, όπου υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλέ διαφορέ. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε βεβαίω είναι να εξετάσουμε αν χρειάζεται περαιτέρω, αν, αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενωσιακής νομοθεσίας για την ε, δίμευση που θα υπερβαίνει τις δυνατότητες που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή η εποπτεία λοιπόν μας δίνει μια καλή βάση για να γίνει αυτή η συζήτηση. Για να είμαι ειλικρινής, η πολιτική μου ομάδα είναι αρκετά επιφυλακτική όσον αφορά την ε, ιδέα να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο εύρος ε, δημεύσεων χωρίς καταδίκη μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίως κατά πόσο είναι υπεύθυνο το να γίνει κάτι τέτοιο, ιδίω εφόσον υπάρχει, ε, υπάρχουν εχέγγυα. Αλλά για μας το καλύτερο εχέγγυο είναι βεβαίως να υπάρχει καταδίκη για να προχωρά κανείς σε κατάσχεση, σε δίμαυση. Και το άρθρο 46 ε, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, για παράδειγμα, μπορεί να απειλείται από τέτοιες πρακτικές. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Περιμένουμε να δούμε και την έκθεση που θα ε, δημοσιευθεί τον Οκτώβριο για την οδηγία του 2002 και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις πληροφορίες και εκείνες που θα ε, περιλαμβάνονται στην έκθεση και αυτές που μας έδωσε σήμερα η Κομισιόν. Κύριε Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Τροπή για Όσον το έγγραφο για της δημόσιας και έχω επαγγελματική προσωπική πείρα και γνωρίζω πόσο αποτελεσματικό είναι για το οργανωμένο έγκλημα αυτό το μέτρο να τους θίξουμε, να τους χτυπήσουμε τα οικονομικά συμφέροντα, να τους αποστερήσουμε από τους πόρους, από τα κέρδη και επίσης θα πρέπει να αποφύγουν να υπάρξει ε, ανάμιξη με την φυσιολογική οικονομία. Οπότε, ακούσαμε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Η ανακρίση είπαμε ότι είναι το 1,1% από το προϊόν εγκλήματος. Και ε, βέβαια, ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η δίμευση χωρίς καταδίκη για την κατόλεμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, όπως ακούσαμε, υπάρχει διαφορά από κράτο σε κράτο τη ρύθμιση. Και βέβαια, ω συνήθω οι μαφίε το εκμεταλλεύονται αυτό για να συνεχίσουν να κάνουν τα δικά τους. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει να θεσπιστεί ο σχετικός ε, κανονισμός ε, που ξεκίνησε τη διαδρομή του το 2018. Ακούσαμε την έκθεση, αναδείχθηκε ο κοινό παρονομαστής, ούτω ώστε να δούμε ποιο είναι το πιο δόκιμο μέσο για να προχωρήσουμε στην ε, νομοθέτηση της δίμευσης χωρίς καταδίκη. Αναφέρθηκε και η τελική εμπειρία όσον αφορά τις δημεύσεις κατά της μαφίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα προς και έτσι να συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα αλλά να έχουμε και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πλεονεκτήμα του Ιταλικού μοντέλου. Έτσι θα πρέπει να δρουν οι δικαστικές αρχές. Να είναι εύστοχη εφαρμογή του μέτρου και από την άλλη μεριά να υπάρχουν όλες οι δικονομικές εγγύησης, όπως υπάρχουν στις συνήθεις ποινικέ διαδικασίες. Και έτσι να δούμε ποια θα είναι τα πιο σημαντικά μέσα, τα πιο αποτελεσματικά μέσα, για να καταπολεμήσουμε το διεθνές διασυνοριακό έγκλημα. περιμένω πώς και πώς το που θα καταλήξει η προσπάθεια της Επιτροπής, θα συμβάλλω και εγώ, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την κοινοτική νομοθεσία ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτση και σας επενθυμίζω λέει ο Πρόεδρος, ότι θα πρέπει να αφήσουμε και κάποιο χρόνο για να συμπληρώσει τα όσα είπε η Επιτροπή. Να υπενθυμίσω απλώ ότι έγινε μια μακρά συζήτηση για τις προτεραιότητε της Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στη διάρκεια αυτής της συζήτηση επισήμανα τη σημασία που έχει η δουλειά μας όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Είμαστε νομοθέτε. Είμαστε νομοθετικό όργανο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα εμείς είμαστε και η κατεξοχή νομοθετική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. διότι εμείς εξαντλούμε και τα όρια της εθνικής κυριαρχίας, γιατί ε, εισερχόμαστε και στα χωράφια του ποινικού δικαίου. Αυτό ακριβώς έγινε και με την οδηγία του 2002, με την οποία εναρμονίστηκαν οι κατασχέσεις χωρίς καταδίκη έπειτα από διαβούλευση των ε, συνομοθετών. Όμω ταυτόχρονα αναθέσαμε στην Κομισιόν και την υποχρέωση να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που αποκομίζονται έπειτα από εγκληματικέ δραστηριότητε και απουσία καταδίκη, δηλαδή προδικαστικά και πριν από την κατάσχεση ποινικέ ή διαδικαστικές διοικητικέ ε, κατασχέσεις, εμπράγματες δηλαδή, όχι κατά προσώπων, αλλά αντικειμένων, περιουσιακών στοιχείων, in rem, κατασχέσεις in rem. Και από αυτή την άποψη σημειώσαμε ότι η ποικιλία προτύπων που προβλέπεται από τις ένομες τάξεις των κρατών μελών δίνουν τη δυνατότητα να αποκομίσουμε ωφέλη σε περίπτωση εναρμόνισης. Και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που πρέπει να λάβει υπόψη της η Διότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν αναδειχθεί μια σειρά από νομικά ερωτήματα στα συνταγματικά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λόγω ακριβώς της ποικιλομορφία και της πολυμορφίας των νομικών κανόνων, όταν προβαίνουν κρατικές αρχές σε δημεύσεις in rem, μέσω νομικών διατάξεων ή διοικητικών αποφάσεων. Τούτου λεχθέντος να ρωτήσω καταρχά την Κομισιόν αν θέλει να σχολιάσει τα όσα ακούστηκαν από τους Ευρωβουλευτές. Έχετε το λόγο και πάλι και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό της της διάταξης. Κύριε Τίγκελ, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το έγγραφο αυτό και για τα ερωτήματα που έχετε θέσει. Να απαντήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου σε κάποια από τα ερωτήματα αυτά. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η απόφαση για το πότε θα εκδοθεί η έκθεση θα ληφθεί από τη νέα ε, Κομισιόν. Θεωρώ όμως ότι εντός του πρώτου ή του δευτέρου εξαμήνου του 2020 είναι ένας στόχος εφικτός. Αλλά όπως είπα θα το αποφασίσει αυτό η νέα Κομισιόν. Το ίδιο ισχύει για όλα τα σχετιζόμενα με προτάσεις νέας νομοθεσίας για το μέλλον. Αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να έχουμε μια πραγματική, ρεαλιστική βάση με στοιχεία η οποία θα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη συζήτηση και στη συνέχεια στην ε, λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά τη χρήση των περισσοκών στοιχείων που κατάσχονται, που δημεύονται, να υπενθυμίσω ότι η ισχύουσα οδηγία 42 περί δίμευσης παροτρύνει τα κράτη-μέλη να εξετάζουν την κοινωνική χρήση αξιοποίηση αυτών των κατασχεθέντων ε, στοιχείων και μάλιστα έχουμε κάνει και μια σχετική μελέτη και διαπιστώσαμε ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν τέτοιο είδους νομικές διατάξεις για την κοινωνική αξιοποίηση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Είναι κάτι που γίνεται, επομένως παρά το γεγονός μάλλον ότι η οδηγία δεν επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικές, απλά παροτρύνει τα κράτη-μέλη να εξετάζουν και αυτή τη δυνατότητα. Να πω επίσης ότι η μεταφορά από τα κράτη-μέλη στο εθνικό, στο εθνικό δίκαιο κατά κανέναν τρόπο δεν ήταν ιδανική. Εμείς μάλιστα έχουμε ήδη ξεκινήσει τρεις διαδικασίες επί παραβάση εναντίον κρατών μελών για τη μη κοινοποίηση ε, της μεταφοράς στο Εθνικό Δίκαιο. Μιλάμε για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο. Είναι υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη. Οπότε ναι, πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά και στη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο από τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια που αφορούσαν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φυσικά κάθε είδος ε, και κάθε μέτρο κατάσχεσης και δίμευσης, χωρίς καταδίκη ιδίω θα πρέπει να σέβεται ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ταυτόχρονα να ε, στραγγαλίζει οικονομικά το, σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Πρόεδρος. Ναι και σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε τις ε, επόμενες κινήσεις της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν. Λοιπόν, Περνάμε τώρα στη μερίσια διάταξη. Ξανά υπενθυμίζω ότι ξεκινάνε οι ψηφοφορίες στις 6. Σε 25 λεπτά περίπου. Και είναι φυσικά η ώρα που θα περιμένουμε πολλούς ευρωβουλευτές οι οποίοι θα προσέλθουν μαζικά, υποψιάζομαι. Επόμενο ε, θέμα, σύστημα φάντο. Επιγραμμικό μητρό Γυνήσεων και ευλαστών εγγράφων. Και κατάργηση τη κοινή δράση του Συμβουλίου 98700 ΔΕΗ. Θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης για το φάντο το οποίο αρχικώς ήταν τμήμα της πρότασης για την Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή και Ακτοφυλακή. Αλλά τελικά Ελήφθη απόφαση να διαχωριστεί έπειτα από αίτημα του Συμβουλίου που εγκρίθηκε και από, το Συμβούλιο των, από τη διάσκεψη των Προέδρων. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μετσόλα που είναι η συγγήτριά μας και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους κοιόδης ε, συντονιστές, ε, εισηγητές μάλλον των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για το επιγραμμικό μητρό γνήσεων και πλαστών εγγράφων. Με αυτό το βήμα θα ολοκληρωθεί και το τελευταίο βήμα για την ε, Ευρωπαϊκή Συνοροφυλική και Ακτοφυλακή. Είχαμε σχεδόν τελειώσει στο τέλος της προηγούμενης ε, ε, κοινοβουλευτικής, κοινοβουλευτικής θητείας. Είναι πραγματικά το τελευταίο μόλις βήμα που πρέπει να γίνει και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαν μαζί μου για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα στο οποίο έχουμε καταλήξει. Η προσέγγιση που έχω υιοθετήσει στην έκθεσή μου για το ΦΑΝΤΟ είναι η βελτίωση, ανάγκη βελτίωση του συστήματο, τη λειτουργία του συστήματο, διευκρινίζοντα ταυτόχρονα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαμόρφωση του ΦΑΝΤΟ. Συγκεκριμένα θεώρησα ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαριστεί τι εννοείται με τον όρο «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Frontex» στο άρθρο 5. Οι τροπολογίες που καταθέτω εξασφαλίζουν ότι το φάντο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για, για την ταυτοποίηση ε, προσώπου που υπάρχουν στο φάντο. Ξανα, επαναλαμβάνω μάλλον, τα δεδομένα του φάντο, οι πληροφορίες του φάντο θα ε, αφορούν μόνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των γνησίων εγγράφων για την καταπολέμηση των πλαστών εγγράφων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της εισήγησής μου, της έκθεσής μου, είναι η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση του ΦΑΝΤΟ. Προτείνω μάλιστα πολλέ από τι εκτελεστικές πράξει που προτείνονται να γίνουν κατεξοδότηση πράξεις γιατί θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται πάντοτε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία ακόμη και όταν η Κομισιόν εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές για το φάντο και τις ε, διαδικασίε ελέγχου και επαλήθευση. Όταν πια θα είμαστε 100% σίγουροι ότι το φάντο λειτουργεί σωστά τότε πιστεύω ότι εκείνοι που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα αυτό θα είναι δευτερεύουσα ε, σημασία θέμα. Γι' αυτό και προτείνω σχετικέ αλλαγέ στα αντίστοιχα άρθρα. άρθρα. Άκουσα και τι ανησυχίε και τι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι συναδελφοί μου από τι πολιτικέ ομάδε όσον αφορά για παράδειγμα το πεδίο ισχύω του κανονισμού που θεωρούν πολλοί ότι είναι υπερβολικά ευρύ. Όμω νομίζω ότι ένα εξαντλητικό κατάλογο εγγράφων δεν θα ήταν ο ενδεδειγμένο τρόπο να προχωρήσουμε. Προτείνω τροπολογίες για τον περιορισμό της χρήσης άλλων επισήμων σχετιζόμενων ε, εγγράφων. Εγγράφων δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν που σχετίζονται με ταξιδιωτικά έγγραφα ή άδεια παραμονής ή ε, έγγραφα ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το έγγραφο πηγή θα προστίθεται κάθε φορά στο φάντο. Έχω λοιπόν υποβάλει και κάποιες ε, τροπολογίες που εξεκαθαρίζουν το ζήτημα και όσον αφορά το Frontex και πρόσθεσα και ένα άρθρο που δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ευθύνες του οργανισμού. Και μία από αυτές τις ευθύνες θα είναι να, να ε, μεταφορτώνει ο οργανισμός όλες τις πληροφορίες που του παρέχουν τα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται ότι οι προφορές που εντάσσονται στο σύστημα θα είναι ομοιόμορφες και συγκρίσιμε. Τέλος, προσπαθώ να εξασφαλίσω ότι ο οργανισμός θα παρέχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο βοήθεια και συνδρομή προς τα κράτη-μέλη όσον αφορά τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων. Ο Frontex ήδη έχει υπερογνωμοσύνη στον τομέα αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να μεγιστοποιήσουν, να εξοπλίσουν στο έπακρο τις δυνατότητες αυτής της εμπειρογνωμοσύνης. Προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση της συνεργασίας μας με τους ε, σκιώδεις εισηγητέ για να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό υπό Φινλανδική Προεδρία, την οποία με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω καθώς και την Κομισιόν για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε κύριε Μετσόλα. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητέ. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Κάλιραντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μένα είναι ένα καινούριο θέμα. Ξεκινώντα λοιπόν, ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που στο προ... στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Και ευχαριστώ και την κυρία Μετσόλα, την εισηγήτρια, για το σχέδιο έκθεση. Μελέτησα τις προτάσεις σας πολύ προσεκτικά και ομολογώ ότι είναι πολύ καλύτερο το κείμενο συγκρινόμενο με αυτό που είχαμε στην ε, πρώτη συνάντηση με την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τους δυο συζητητές. Δεν αμφισβητώ τη σημασία του θέματος. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με το σύστημα αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάποιες ανησυχίες παραμένουν. Δεν θα μιλήσω για προτάσεις για τη σύνταξη του κειμένου, θα υποβάλω τις σχετικές προτάσεις, αλλά θέλω να τονίσω κάποια σημεία. Ένα σημείο που αναφέρετε κι εσείς είναι το θέμα του κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα. Εφόσον είναι μια βάση δεδομένων, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Βέβαια, η συγγήτρια έχει βάλει κάποιες ιδέες για ελαχιστοποίηση των δεδομένων και ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Παρόλα αυτά, πρέπει να είναι σαφέστερη η, ε, η δήλωσή μας να εκφράζουμε σαφώς ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Δεύτερη ανησυχία για τα σημεία πρόσβασης. Αναγνωρίζω τις προσπαθειές σας και η, γενική εικόνα είναι καλύτερη. Υπάρχουν όμως τόσα διαφορετικά επίπεδα και τόσα πολλά σημεία πρόσβασης που πρέπει να το κάνουμε σαφέστερο. Χρειάζεται ακόμη λίγο δουλειά εδώ. Τέλος, ένα θέμα για τα έγγραφα ο μη πλήρης κατάλογος σας διαβεβαιώνω ότι τα κράτη-μέλη εκατοντάδες επίσημα έγγραφα μπορούν να εκδίδουν. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε ένα περιορισμένο κατάλογο επισήμων εγγράφων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια ως προς το τι πρέπει να παρέχουν τα κράτη-μέλη. Αυτά και θα είμαι στη διάθεσή σας, ε, κυρία Συγήτρια. Προσβλέπω στη συνεργασία μας. Ωραία. Ο κύριος Τουντοράτσε, εκ μέρους της Renew Europe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ρομπέρτα Μετσόλα για την εξαιρετική αυτή, για το πρώτο αυτό σχέδιο έκθεσης. Όπως είπε και η συνάδελφος, και εγώ πιστεύω ότι η έκθεση υπογραμμίζει κάποια από τα στοιχεία που αποτελούσαν ανησυχίες και για μας. Το δεύτερο είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογής. Το πρώτο σχέδιο πρότασης υπήρχε ορισμός ε, του Φάντο και η άμεση αναφορά ε, σε αυτά τα οποία ε, αποθηκεύει ήδη το Φάντο δείγματα εγγράφων. Δηλαδή, ε, είναι μια καλή τροποποίηση και όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και για μας είναι σημαντική ανησυχία, δεν είναι σαφές το τι αποθηκεύεται στο σύστημα αυτό και αυτό μας δημιουργεί μια αμφιβολία για το τι ρυθμίσεις θα χρειαστούν όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα και η συγγήτρια είπε ότι πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και αυτό μας βοηθά με τον περιορισμό των χρήσεων για τα προσωπικά δεδομένα. Υποστηρίζω λοιπόν αυτή την τροποποίηση. Τέλος, η τροπολογία 80 δέλτα χωρίς να θέλω να μιλήσω τώρα για τη σύνταξη, ε, σχετικά με τις υποχρεώσεις του οργανισμού, βρίσκω τις ε, τροποποιήσεις χρήσιμες. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που τροφοδοτούν το σύστημα και των τρίτων μερών, όπως αεροπορικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη ή άλλοι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ε, ε, αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπρικμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Μετσόλα, για την δουλειά που έχετε κάνει. Ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής. Σε πολλά σημεία διείσταται η άποψή μας από τις απόψεις του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, για τη σύνταξη. Παραμένει κάποιο ερωτηματικό για τη βάση δεδομένων την οποία έχουμε δώσει στη Frontex ε, αντί στην ε, Europol, κυρίως διότι η Europol είναι υπεύθυνη για την αστυνομική συνεργασία. Ακούσαμε τα επιχειρήματα του Συμβουλίου για την νομική βάση. Παρόλα αυτά, μας ενδιαφέρει το πώς θα εξελιχθεί το θέμα και όταν ε, μεταφέρονται αρμοδιότητες από τον ένα οργανισμό στον άλλον και ιδιαίτερα προς τον Frontex. ανέφερε η συνάδελφο στο θέμα των προσωπικών δεδομένων. Θέλουμε να αναφέρεται ρητά ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα. Θέλουμε λοιπόν μια σχετική τροπολογία. Και θέλουμε να έχουμε εγγύησει και διευκρινήσεις για τα επίπεδα πρόσβασης στη βάση δεδομένων. και θα πρέπει να διευκρινιστεί και το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Ταρντίνο μετά τους πρασίνους, του ID. Ευχαριστούμε την κυρία Μετσόλη για όσα έκανε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η αφετηρία. Πολύ καινοτομή πρόταση της κυρίας Μετσόλα Παρ' όλα αυτά επιφυλάσσουμε να δούμε εις βάθος, γιατί στο παρελθόν υπήρχε θέμα με το Frontex και το σύστημα Φάντο. Είναι σημαντικό το θέμα του, της διάκρισης με τις εκτελεστικές πράξεις και της ε, ε, πράξης. Είναι αυτά τεχνικά ζητήματα και θα πρέπει να ξαναδούμε την τροπολογία 32. Επαναλαμβάνω πάντως ότι το κείμενο είναι μια πολύ θετική αφετηρία. Ο κύριος Μπουσαντέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, βεβαίως να ευχαριστήσω πρώτα την εισηγήτρια για τη δουλειά της τελευταίες εβδομάδες για να δούμε πώς θα τροποποιηθεί αυτή η πρόταση που συζητούμε. θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν υποχρεούνται ή όχι τα κράτη-μέλη να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες για το φάντο. Αν ναι, το κράτος μέλος θα ορίσει ποια υπηρεσία του θα κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται για τις τεχνικές προδιαγραφές, τι γίνεται για την αποθήκευση των δεδομένων, πώς θα ελέγχονται οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί, πώς θα επιβιώνονται. Ναι, το, το ξεκαθάρισε η Επιτροπή, αλλά δεν ξέρω τι είναι με τις οι πράξεις. Θα πρέπει και κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει πιο σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο. Γιατί έτσι όπως τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για κάποια πολύ τεχνικά θέματα. Πότε θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι να προστατευτεί και η Frontex και η τεχνική. Επίσης, περιορισμένη πρόσβαση για κάποια διαβαθμισμένα έγγραφα, τα οποία είναι αντικείμενο δικαστικής έρευνας. Άρα, να κάνουμε ό,τι γίνεται, ούτως ώστε να διευκολύνουμε δικαστές και αστυνομικούς. Πιστεύω ότι με την κοινή προσπάθεια θα καταλήξουμε σε συμφωνία και θα μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε και τώρα για την ΚΟΕ. Έχουμε δύο σκιώδες, την κυρία Ρέντ, δεν τη βλέπω, δεν είναι εδώ. Ο κύριος Καστάλντα. Άρα δεν έχουμε κάποιον από την ΚΟΕ να μας πούν τη γνώμη τους για την κυρία Ε, τότε, εν αυτή τη, περιπτώση, ξαναγυρίζουμε στην κυρία Μετσόλα. Η Ε, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Όλους που μίλησαν με θετικό πνεύμα, αισιόδοξα, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά ό,τι ακούστηκε θα το λάβω υπόψη. Και θα ενημερώσω όλους τους εμπλεκόμενους και να έχουμε, θα φροντίζω όσο γίνεται περισσότερο χρόνο τόσο ώστε όλοι να εξηγηθούν το κείμενο. Να έχουν όσο χρόνο θέλετε για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι αποδεκτό από όλους. Ευχαριστούμε κύριε Μητσολογία για το κείμενό σας και τη δουλειά σας. Υπάρχει συνένεση όσον αφορά το κείμενό σας. Οι τροπολογίες έχουν προθεσμία την 15η Οκτωβρίου, Οπότε ολοκληρώσουμε για αυτό το σημείο της και θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Έξι ώρα προβλέπεται η αρχή της ψηφορίας, άρα έχουμε λίγα λεπτά και γι' αυτό και σας προτείνω μια πολύ πολύ μικρή διακοπή. Πρέπει να έχετε όλη την ηλεκτρονική σας κάρτα για την ψηφορία. Σε λίγα λεπτά αρχίζουμε. we go. Now we go. Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω. Κάποιοι από εμάς ήμασταν εδώ όλη μέρα. Ξεκινήσαμε με την ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ στις 9 το πρωί, μετά συνεχίσαμε στις 2.30 και σχεδόν 4 ώρες μετά να είμαστε και πάλι εδώ και περνάμε στα τελευταία σημεία της διάταξη διάταξης, στις ψηφοφορίες δηλαδή. Και μάλιστα παρέτεινα όσο μπορούσα την ψηφοφορία, προκειμένου όσοι είχαν ξεχάσει την ηλεκτρονική τους κάρτα να την αποκτήσουν, να τους τη φέρει κάποιος, για να εξασφαλίσουμε επίσης ότι εκπροσωπούνται επαρκώς και με τον προβλεπόμενο τρόπο όλες οι πολιτικές ομάδες. Αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ανακοινώσω όμως ότι έχουμε μπροστά μας 10 ψηφοφορίες διαδοχικές. 10 τον αριθμό. Λίγο ως πολύ πρόκειται για ζητήματα εκκρεμούντα από την προηγούμενη θητεία. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στην τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελήφθη απόφαση από τη συνεδρίαση των συντονιστών που είναι το αρμόδιο όργανο ότι η Κομισιόν δεν θα χρειαστεί, δεν θα πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση, να λάβει νέα πρωτοβουλία για, τον κάθε, για το κάθε θέμα. Αποφασίσαμε να αναλάβουμε ξανά αυτά τα ζητήματα που εκκρεμούσαν από την προηγούμενη θητεία και να τα προχωρήσουμε. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο του 71 του εσωτερικού κανονισμού, χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα προαγάγουμε τα θέματα που είχαμε ολοκληρώσει σε πρώτη ανάγνωση στην προηγούμενη θητεία. Στην ουσία δηλαδή ψηφίζουμε για την έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς να χρειάζεται επιτροπή συνδιαλλαγής. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία. Ιδίω για εκείνου που είστε νέοι στην Επιτροπή ΛΥΜΠ σημαίνει ότι χρειαζόμαστε από τα 68 τακτικά μέλη, χρειαζόμαστε 35 ψήφους θετικές υπέρ για να προαγάγουμε τους φακέλους αυτούς και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει. Γι' αυτό και ήθελα να εκπροσωπούνται επαρκώς όλες οι πολιτικές ομάδες. 30 ψήφοι υπέρ χρειάζονται. Λοιπόν, ξεκινάμε τι ψηφοφορίε. Με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων σε εσωτερικά σύνορα. Ψηφίζουμε επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. έκθεση Τάνια Φαγιών και ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. We, we had a problem with Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τους σοσιαλιστές. Έχουμε έναν υπεράριθμο από τους σοσιαλιστές. Όχι πια, ωραία, λύθηκε το πρόβλημα. Άρα, ολοκληρώνει η ψηφοφορία. Πέρας, 43 υπέρ, 43 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, 12, 12 ε, κατά, 11 αποχές. Εγκρίνεται. Κανονισμός VIS. Η συζήτηση είναι ο συνάδελφος Παύλο Ρανζέλ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Θετικό το αποτέλεσμα, 53 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 8 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ρανζέλ, συγχαρητήρια και κυρία Ταγιών. Φαγιών. Ενισχυμένη πλειοψηφία. Θέσπιση προγραμμάτων ανταλλαγών συνδρομή και κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κυβδηλία για την περίοδο. Όχι, όχι, όχι. Έκανα λάθο. Με συγχωρείτε. Πήγα στον Περικλή, αλλά δεν ήταν αυτό. Ξέχασα τι κοινοτικέ στατιστικέ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Η είναι ο κύριο Ότκιν. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά με την κάρτα σα. Πέρα τη ψηφοφορία. Ναι, πέρασε. Με μεγάλη και ενισχυμένη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα περνάμε στον Περικλή. Στο πρόγραμμα Περίκλες 4. Κλέρ Ντέιλι είναι η εισηγήτριά μας. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Θέσπιση του προγράμματος Δικαιώματα και Αξίες. Ένα από τα θέματα που σχετίζονται με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η συγγήτρια είναι η κυρία Άλλη Κούνκε. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ με την κάρτα σας. Πέρα τη ψηφοφορίας. Επίσης εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Θέσπιση τομείου Ασύλου και Μετανάστευση. Επίση, θέμα που σχετίζεται με το ΠΔΠ. Η συγκίτρια είναι η κυρία Μίριαμ Ντάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Εγκρίνεται, εγκρίνεται και αυτό. Επόμενο σημείο. Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτική στήριξη για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων. Η και πάλι κυρία Τάνια Φαγιών. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τώρα. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται συγχαρητήρια και πάλι. Με ενισχυμένη πλειοψηφία. Επόμενο θέμα θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η συγγήτρια κυρία Μόνικα Χολμάια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ενισχυμένη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Χολμάια. Πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Εισηγητής είναι ο Πάτρικ Γιάκη. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια και πάλι. Και περνάμε στο δέκατο σημείο κατάλογος κρατών των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να κατέχουν θεώρηση και εκείνων που εξαιρούνται, συγκεκριμένα Κόσοβο. Και πάλι εδώ η συγκήτρια κυρία Φαγιών, ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ, άρχιτη η ψηφοφορία, τους της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους τους συγητές και τις συγητρίες για την προαγωγή των θεμάτων αυτών για να περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Καλό βράδυ σε όλους και σας ευχαριστώ. Γεια σας.